Tu Γεια σας κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Καλωσορίσατε ορίσατε σε όλους, σε όλες. Στο, στο πρώτο τμήμα τη συνεδρίασή μας αντικαθιστώ την κυρία Βαζολή. Δεν βρίσκεται εδώ, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίζει αυτή τη στιγμή στι Βρυξέλλες αλλά σε άλλο χώρο. Η πρόεδρος κυρία Ζολή θα έρθει πιο αργά το απόγευμα. Αφετέρου, η διερμηνία, η γενική, η γενική διερμηνία, η γενική διαρμηνία δεν ήταν δυνατόν να μας δώσει διερμηνία από τα Σουηδικά και προς τα Σουηδικά. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο παραλείπω αυτά και θέτω σε έγκριση την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Λαμπρά. Υιοθετείτε συνεπώς και έχετε επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της 18 Οκτωβρίου ενεστώτος. Εν υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά αυτά τα πρακτικά. Παρακαλώ, παρακαλώ να το υποβάλλετε στο στη γραμματεία πριν από το πέρας της συνεδρίασης. Διαφορετικά θα υιοθετηθεί αυτομάτως εφόσον δεν υπάρξουν δικά συνδείξεις. Τώρα, ανακοινώσεις της Προεδρίου. Δεν έχω να κάνω. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεν είχαμε ερωτήσει τις οποίες έπρεπε να θέσουμε προς την Κομισιόν για τη συνεδρίαση, άρα περνάω και το πέμπτο σημείο της ημερήσιας, τέταρτο σημείο. Όσον αφορά την Κομισιόν αυτή καθεαυτή, μήπως υπάρχει καμία αναγγελία εκ μέρους ή ανακοίνωση εκ μέρους της Κομισιόν. Φαίνεται πως όχι. Νομίζω πως η συνεδρίαση θα πάει πολύ γρήγορα. Είναι Δευτέρα και θα τελει... περατώσουμε εντάχει. Ερχόμεθα λοιπόν στο επόμενο. Χρηματοδότηση της καινοτομίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς η Οικονομική Επιτροπή εκπονεί μια έκθεση όσον αφορά αυτή την καινοτόμο χρηματοδότηση, μάλλον τη χρηματοδότηση καινοτομίας. Εμεί είμαστε λοιπόν μια επιτροπή που θα δώσουμε την άποψή μα σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού. Το κείμενο έχει σαν στόχο τρει τομεί, το δημοσιονομικό, το εναλλαγή του κλίματος και την ανάπτυξη. Η επίδραση τη κλιματική αλλαγή. όσον αφορά την ανάπτυξη αφορά ιδιαίτερα δική μα επιτροπή η οποία Εφάνει ότι ήταν πολύ δραστηρή σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη της χρηματοδότησης, καινοτόμα χρηματοδότηση, Νομίζω πω άπτεται και αυτό του τομέα του δικού μα και της Επιτροπή μας. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντεβά, ο οποίο ορίστηκε εισηγητή επί του θέματος αυτού. Κύριε Ντεβά, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κοιτάζοντα ακόμη και αυτή την έκθεση όσον αφορά την χρηματοδότηση καινοτομία. Εδώ στην Επιτροπή μας μας δίνει τη δυνατότητα να κατέβουμε τον ίδιο κατήφορο, να φύγουμε από την ίδια σκέψη και τον τρόπο σκέψης που είχαμε εδώ τα και τελευταία χρόνια σε αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο επ' αυτού και να διαρωτηθούμε κατά πόσον υπάρχουν άλλοι τρόποι για καινοτόμα χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τι αναπτυσσόμενε χώρε αλλά και τον φορολογούμενο μα. Κοιτάζω σε αυτή την έκθεση λοιπόν, σαν έκθεση, σαν ε, επιφορτισμό να δώσω την, τη γνωμοδότηση, βλέπω πραγματικά πως η οικονομία χάνει πάρα πολύ χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, έγιναν περικοπές 25% του προϋπολογισμού το ίδιο έγινε το αυτό σε άλλε χώρε της ΕΕ. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για χρηματοδότηση καινοτομία, θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε στους παλιέ παλιές μεθόδους ναι, συλλογή χρημάτων αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να βρούμε, όχι με το παρελθόν, όπως γίνεται στην Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο αυτή τη στιγμή να πυρκόπτει ο προπολογισμός κατά 25 και 30%, κατά αυτόν τον τρόπο που έγινε βέβαια αυξήθηκε πάρα πολύ η φορολόγηση των ε, εγκλέζων φορολογουμένων. Έτσι λοιπόν πιστεύω έχουμε μια επιλογή που είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Θα πρέπει να πούμε στους φορολογούμενους μας αυτή τη στιγμή ότι είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε νέες προοπτικές. Αλλά είναι αυτό ότι θα πρέπει να έχουμε πάντοτε αυτή την υπόσχεση που έχουμε κατά νου δώσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις, κοινο... τις καινοτομίες κατά 25% για να φτάσουμε τους στόχους. Επειδή όμως αυτό το πράγμα το οποίο θα έχουμε θέσει και δεν το έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι στιγμή, ούτε ακόμα και στις ΗΠΑ, αυτό οδηγεί πραγματικά προς την παινία. Το να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να ξεπατώσουμε την παινία δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή με αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό που θα, για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα μιας αηφόρας προσπάθειας η οποία γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ο γι' αυτό είναι ο για τον οποίο θα πω, ήθελα να πω ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες θα είναι δίκαιες σωστές για αυτούς οι οποίοι δέχονται τα χρήματα αυτή, αυτά και σαν εταίροι εμείς αυτή τη σχέση που έχουμε μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσομένων χωρών. Δεδομένου ότι, ότι πολύ περισσότερα χρήματα, ότι τεράστια χρήματα, φρέσκο χρήμα χρειάζεται και θα πρέπει να ευρεθεί αυτό το χρήμα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις οι οποίες ε, σε μια, αλλαγή, ε, σε μια εποχή τέτοιων αλλαγών οι οποίες υπάρχουν. Χρήματα για τα οποία θα πρέπει να δοθούν ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να μειώσουν και να φτάσουν πραγματικά σε εκείνο το σημείο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και νομίζω πως 100 ε, εκατομμύρια λέγεται. Δεν είναι χρήματα, γιατί έχουμε μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή να δώσουμε αυτό το, το ποσό. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσει, υπάρχουν πιέσει οι οποίε ασκούνται, Ανθρώπινε αφετέρου υπάρχουν προσδοκίε, οι οποίοι, προσδοκίες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν αυτή τη στιγμή να προστατεύσουν τον πλανήτη, να μειώσουν αυτές τις επιπτώσεις που υπάρχουν από τον πλανήτη, Δεδομένου αυτών των προστοκιών των ανθρώπων να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους το 2015, το 2015 οι αγαπησόμενες χώρες είναι εταίροι μας τι θα πρέπει να κάνουμε με όλα αυτά, μια κοινή τέρημα; εάν πραγματικά δώσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο σκέφτηκα πώ μπορούμε εμεί αυτή τη στιγμή να έχουμε με νέε ιδέε, νέου τρόπου για να τους βοηθήσουμε για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και αυτές τις προκλήσεις που έχουμε. Ένα πράγμα το οποίο βλέπω στην έκθεση την οποία σας καταθέτω είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εάν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή πραγματικά στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς εμείς εδώ συνεδριάζουμε και μιλάμε η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα και οι αναπτυσσόμενες χώρες χρένουν 100 δις το χρόνο εάν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει βοήθεια 60 ε, από την έψη και το υπόλοιπο, το, υπόλοιπο από το υπόλοιπο του χρόνου. Αν αυτό όμως συμβεί 800 δις ευρώ μπορούν να αποκτηθούν χάρη σε αυτή την επένδυση που έχει γίνει. Και αυτό δεν αποτελεί μέλος της, επίση, μέλος της ε, οικονομίας, δεν είναι μέλος της, του ΑΕΠ δεν είναι μέρος καν. Αυτά τα 800 δις έρχονται, προέρχονται από αυτές και όπως το εξήγησε η συνάδελφός μου πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε εταιρείε και σε κέντρα offshore. Αυτά τα ποσά δεν δημιουργούν βεβαίω πλούτο και δεν αναπτύσσουν τι αναπτυσσόμενε χώρε δεν καταπολεμάνε την παινία, τη φτώχεια. κύριος είδε που πάνε αυτά τα χρήματα, αλλά πηγαίνουν ασφαλώ. σε παραδείσου, φορολογικούς παραδείσου, στην Καραϊβική και αλλού, για έτερους σκοπούς, αλλά όχι, εν πάση περιπτώσει, για την ανάπτυξη των, φτωχών, των αναπτυσσομένων χωρών. Αν υποτεθεί ότι μπορούμε να έρθουμε αυτή τη στιγμή με μηχανισμούς που μπορούμε να σταματήσουμε αυτά τα χρήματα να φεύγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αν υποθέσουμε από την άλλη ότι έχουμε αυτά τα 800 δις και να είναι η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στις βοήθειες σε αυτές τις χώρες και ότι μπορούμε να τα εισάγουμε ε, εκ νέου αυτά τα λεφτά στην Επιτροπή, στις χώρες αυτές να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα, να διατηρηθούν αυτά για περαιτέρω ανάπτυξη, να δημιουργήσουν πλούτο σε αυτές τις χώρες και βοήθεια κλπ. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι αν σταματήσουμε αυτά τα χρήματα να λελατούνται από αυτές τις χώρες και διακριρήσουμε αυτά τα χρήματα, αυτά τα ποσά μέσα στη χώρα, θα υπάρχει μια τεράστια διαφορά τα οποία θα γίνει, ιδιαίτερα εις όφελος, προς όφελος των φτωχών ανθρώπων της περιοχής αυτή εάν τα χρησιμοποιήσουμε οκτώ φορές πάνω από το ποσό που της βοήθειας το οποίο δίδεται δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, νέα γεωργία, νέα βιομηχανία, τα πάντα, κτηνοτροφία τα πάντα. Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής, πώς μπορούμε να διατηρηθεί αυτό το χρήμα να μην πηγαίνει, πώς μπορούμε να το εμποδίσουμε να πηγαίνει στους φορολογικούς παραδείσους. Πώς μπορεί το χρήμα να χρησιμοποιηθεί επιτόπου. Πώς μπορούμε αυτές οι ροές να διατηρηθούν, να παραμείνουν εκεί που πρέπει να γίνουν. Μιλάμε για, την, για το φόρο, τόμπιν κλπ. Αλλά θα πρέπει να διαρωτηθούμε μια απλή ερώτηση πώς μπορούμε ήδη πέρα από αυτό το τόπι να διατηρηθούν αυτά τα ποσά εκεί, να μην φεύγουν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς κατά αυτόν τον τρόπο όπως ώστε το, το χρήμα αυτό να μην ανακυκλώνεται προς τα έξω. Εάν το κατορθώσουμε αυτό, τότε εμείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά τα που αποσχεθήκαμε στο Κινικόλ θα μπορούμε να έχουμε ένα εταιρικό σχήμα ε, με καλή διακυβέρνηση, με διαφάνιση και με αμοιβαία υποστήριξη ένθεν και κήθεν το οποίο θα δεσμεύσει τον καλύτερο κόσμο, τα καλύτερα μυαλά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, καθώ επίση και αυτού του ανθρώπου που κατέχουν αυτό το κεφάλαιο και το οποίο το εκραίουν από αυτέ τι χώρε. Θα είναι ένας, ένα νέο partnership, ένα νέο εταιρισμό, ένα νέο τρόπο αντιμετώπιση και σκέψη. Αυτή μπορεί να είναι η λύση για τα θέματα αυτά τα οποία Αυτό το οποίο λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε είναι είναι πώς θα εμποδίσουμε αυτά τα λεφτά. Αν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα διασώσουμε και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, θα βοηθήσουμε Επίση, πάρα πολύ το θέμα της κλιματικής αλλαγής διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει περισσότερη ροή, θα υπάρχει περισσότερη ε, ρευστότητα στι χώρε αυτές εφόσον εμποδίσουμε να φεύγει αυτό το χρήμα να εξάγεται από αυτές τις χώρες. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε αυτούς όλους οι οποίοι θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις τράπεζές τους κλπ, να δημιουργήσουν προγράμματα δημιουργίας θέσεων, θέσεων εργασίας κλπ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν για καλή διαχείριση, για, για, για τη διακυβέρνηση, για τις τράπεζες, για τη διοίκηση, για χρηστή διοίκηση κλπ. Ούτως ώστε αυτά τα χρήματα να μην βγαίνουν παράνομα από τις χώρες αυτές, να μην δημιουργούν να δημιουργήσουμε μια partnership, μια εταιρισμό νομικό, δικαϊκό, ο οποίος θα προστατεύει τους πολίτες αυτών των χωρών και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν τα παλαιότερα χρήματα τα οποία υπάρχουν για την ανάπτυξή τους. Αυτό είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να τους προσφέρουμε καθότι γνωρίζουμε και γνωρίζουμε καλά ότι οι ηγέτες αυτών των χωρών, οι ηγέτες και αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή παίρνουν αυτά τα λεφτά, τα λελατούν στην κυριολεξία αυτά τα λεφτά γιατί δεν, υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχει νομικό συστός, υποδομή, δεν υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση κλπ. κλπ. Το έχουμε τα παραδείγματα από αυτή τη χώρα. Πήγαμε στο Κατμαντού και είδαμε ότι είδαμε την επιτροπή κοινή του, όπου το, το κοινοβούλιο του Νεπάλ κοίταζε αυτή τη στιγμή πώς διακυβερνά τη χώρα και πώς γίνεται η κυβέρνηση της χώρας αυτής. Βεβαίως θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί, οι, στο που πήρα για παράδειγμα, να βοηθηθούν αυτοί οι περισσότεροι για να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη, για να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός προς τις αρχές, προς το δίκαιο και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα περιγράφουμε στην έκθεσή μου και σας ευχαριστώ πολύ. Okay, merci, monsieur... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντεμπά θα σα ρωτήσω τώρα. Θα ξεκινήσω τον κύριο Γκερέρο. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Γκερέρο. Γιατί δεν πρέπει να καθυστερήσουν περαιτέρω. Ο κύριος Γκερέρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντέβα. Περισσότερο για την παρέμβαση, την προφορική του παρέμβαση που ήταν πολύ πιο εκτεταμένη από την ίδια του την εισήγηση. Κάλυψε πολλά ζητήματα τα οποία περιέχονται στον τίτλο της εισήγησης. Νομίζω ότι εστιάζει ε, πολύ σωστά. Υπό την έννοια ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια συμπεριλαμβανομένων και νέων πηγών χρηματοδότηση, δεν μπορεί να λύσει από μόνη τη το πρόβλημα τη φτώχεια. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε επίση ότι αν δεν διατηρήσουμε την προσήλωσή μα και την δέσμευσή μα σε αυτή την ε, αναπτυξιακή βοήθεια με νέε πηγέ χρηματοδότηση, σίγουρα θα μείνουμε ακόμα πιο μακριά από την εκρήωση τη φτώχεια. Γιατί η φτώχεια μειώνεται με συνεπεί πολιτικέ και με μια σειρά άλλων δράσεων στι οποίε αναφέρθηκε ο κύριος Ντέβα. Συνεπώς συμμεριζόμαστε αυτό το σημείο και το, το θέμα της ε, καταπολέμησης ε, των ε, παράνομων ροών κεφαλαίων, την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, προστατεύοντας τι αναπτυσσόμενε χώρες και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε ε, να βοηθήσει έτσι ώστε να συναυθεί μια παγκόσμια συμφωνία ανταλλαγής ε, χρηματοοικονομικών στοιχείων τέτοιου τύπου ε, με συγκεκριμένε κυρώσεις μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως η έκθεση της Επιτροπής ΕΚΟΝ αφορά καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης Λοιπόν, ω σκιώδη συγητή των σοσιαλιστών θα ήθελα η έκθεση του κ. Ντέβα να ασχοληθεί και με ορισμένου από αυτού του μηχανισμού χρηματοδότηση, οι οποίοι συζητώνται και έχουν συζητηθεί στο παρελθόν στην Επιτροπή μα. Και επί των οποίων συμφωνήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, ε, ο φόρο επί των διεθνών ε, συναλλαγών. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς διεθνή συμφωνία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί τέτοιου είδους φόρος. Όμως, ακόμα και η ίδια η Κομισιόν έχει θέσει το θέμα της εισαγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός τέτοιου φόρου. Επίσης, φόροι επί των μεταφορών. Υπό την έννοια ότι ε, αποτελούν αντικίνητρο στη χρήση άνθρακα και μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Επίσης θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος των εμβασμάτων που στέλνουν οι μετανάστες ε, στη χώρα προελευσής τους. γιατί μου ζητήσατε πρόεδρε να είμαι σύντομο, θα σταματήσω εδώ. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι θα αποστείλω στον κύριο Ντέβα ορισμένε τροπολογίε, ε, οι οποίε δεν έχουν σχέση τόσο πολύ με την ουσία. Όχι, γιατί ασφαλώ χρειάζονται καινούργιε οδοί, καινούργιοι τρόποι. Ε, πλην όμω με τι τροπολογίε αυτέ που θα προτείνω θα αναφερθώ σε καινοτόμε ε, λύσει χρηματοδότηση, μια και το θέμα αυτό ακριβώ είναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Στο έργο της ε, ε, Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Ο λόγος του κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ Νέρτζ για, για την έκθεσή σου για ορισμένες πολύ εξαιρετικές θα έλεγα προτάσεις που έχει υποβάλει. Θέλω να σχολιάσω κάποια θέματα. Ε, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια αποτελεί ταυτόχρονα και επένδυση σε αυτές τις χώρες. Ε, χρειάζονται ε, χρειάζεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ε, να θεωρηθεί και ως κομμάτι των επενδύσεων που κάνουν σε αυτέ τι χώρε. Και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τι ευάλωτε οικονομίε του είναι η μείωση του κόστου ε, των εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι χώρε αυτέ. Γιατί όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα εμβάσματα είναι πολύ μεγαλύτερα σε όγκο, σε ποσό από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια την οποία χορηγούμε προς αυτές τις χώρες. Ε, δεν διαφωνώ για αυτά που είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το 0,7% του ε, ε, ε ως αξιακή βοήθεια. Το Σεπτέμβρη, στην Σύνοδο Κορυφής των Στόχων της Χιλιετίας μάλιστα, έγινε, αναλύθηκε η δέσμευση ε, να ε, υιοθετηθεί ένας φόρος επί των ε, συναλλαγών, οικονομικών συναλλαγών. Συνεπώς ελπίζω και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και με την ευκαιρία του καφέ που μας σερβίρεται σκέφτομαι το εξή. Έχουμε τα διάφορα εμπορεύματα όπως ζάχαρη, κακάο, καφές κλπ. που σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον ανεξόμενο κόσμο. Τα αγοράζουμε σε μια συγκεκριμένη τιμή και τα εμπορευόμαστε μέσω ε, ε, αγορών στις ε, οποίες η τιμή αυξάνεται μέσω των διαφόρων μεσαζόντων. Όμως αυτή η αύξηση δεν επιστρέφει ούτε ως ποσοστό στους παραγωγούς. Ε, μην ξεχνάμε ότι πολλές φορέ φορολογείται αυτή η προσθέμενη αξία. Κανένας από αυτούς τους να δεν επιστρέφει όμως στο, στους παραγωγούς. Ίσως θα έπρεπε ένα κομμάτι να σημαίνει αυτό. Επίσης, για την εξωτερική βιομηχανία χρειαζόμαστε ένα φόρο ενδεχομένως. Ε, μιλάμε για, όχι μόνο για πετρέλαιο και για χαλκό, μαγνήσιο και πολλά άλλα ε, υλικά τα οποία εξορίσσονται, μέταλλα κλπ. Ε, είναι σημαντικό όταν γίνεται εξόριξη από αυτές τις χώρες να πληρώνεται ένας φόρος που θα καταλήξει σε αυτές τις χώρες πάλι. Και πάνω από όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά. Είναι σημαντικό να κλείσουν οι φορολογικοί, offshore φορολογικοί παράδεισοι, διότι εκεί γνωρίζουμε πως πολλές ε, ε πολυεθνικές εταιρείες ε, που είναι κατεστημένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους, επαναλαμβάνω, για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. Το κλειδί όμως για όλα αυτά είναι η διαφάνεια ε, χρηματικών ροών σε όλο τον κόσμο. Γιατί μόνο με αυτόν τον ε, τρόπο υπάρχει εξασφαλίζεται λογοδοσία και γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Λόγω στον κύριο Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο Ντεβά. Διότι η εισαγωγή του ήταν πολύ σοφή, ε, χαρακτηρίζεται από κοινή λογική. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις στα εισαγωγικά του σχόλια. Σε ό,τι αφορά τη λαιλασία των, ε, ε, του πλούτου ε, στις αντισόμενες χώρες, ασφαλώς και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω αν πρόκειται για 800 δισεκατομμύρια. Ποτέ δεν θα το μάθουμε, όπως δεν ξέρουμε πόσα, ποια ποσά ξεφεύγουν από τους δικούς μας εφόρους στις δικές μας φορολογικές υπηρεσίες. Ακόμα και με τους μηχανισμούς που διαθέτουμε δεν έχουμε καταφέρει εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά ταυτόχρονα και με τριόφρονες για το κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Τώρα, τι σημαίνει καινοτόμος χρηματοδότηση. Σημαίνει πολλαπλησιασμό των πόρων ή να ε, καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερε τι αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς να φτάσουμε στο 0,7%. Αν είναι αυτό, έχω κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν θα πρέπει να ε, οδηγήσουμε τον αναγνώστη σε παραπλάνηση. Δηλαδή, θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο ε, του, της, ε, ε Ευρωπαϊκής Συμφωνίας του 2005. Και Αυτό, αυτή η Ευρωπαϊκή Συνένεση Ανάπτυξης του 2005 ε, ε, θα πρέπει να κάνει σεβαστό το 0,7%. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς και θα πρέπει το Συμβούλιο, τα κρατημέλη δηλαδή, να μας πούν τι σκοπεύουν να κάνουν. Διότι αν ένα κράτος μέλος ε, παραβεί τη δεσμευσή του, θα αποτύχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και έχει επαναλάβει πολλές φορές. <clears throat> Θα πρέπει να το πούμε αυτό στο Συμβούλιο ακόμα και αν το Συμβούλιο κοφεύσει. Θα το πω και παρουσία της κυρίας Άστον σε λίγο. Τρίτον, Θα πρέπει να ξεκινήσουμε προβληματισμό σε ό,τι αφορά την στρατηγική που θα μπορούσε να συνδυάσει τις επιθυμίες του κ. Ντέβα με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε δηλαδή ε, να ε, δημιουργηθεί ένας διάλογος ε, μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, ή κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών που των οποίων οι χώρες λαιλατούνται, των οποίων οι φυσικοί πόροι λαιλατούνται, υπάρχουν άπειροι τρόποι να γίνουν αυτοί οι λαιλατήση. Για παράδειγμα, ε, να εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο αυτό χωρίς να πληρώνουμε τις ε, δίκαιες τιμές ή μέσω ε, σκοτεινών δρόμων κλπ. Υπάρχουν, υπάρχει πάντοτε παραθυράκια. Υπάρχουν πάντοτε παραθυράκια. Αυτό το βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν διάφορες ε, τέτοιες ε, απόπειρες, επιτυχημένες απόπειρες φοροδιαφυγής, μαύρης οικονομίας κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νταβός όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να μπορέσουν να προβληματιστούν και οι επιχειρήσει που εργάζονται σε αυτές τις χώρες και οι δικαιούχοι τη βοήθειας και οι δωρητέ κλπ. Διότι οι επιχειρήσει είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετάσχουν ε, διότι δεν είναι υποχρέωσή μόνο να τηρούν τη δική μα νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την νομοθεσία των χωρών στι οποίε ε, ε, δραστηριοποιούνται. Λοιπόν, έχουμε κανόνες και θα πρέπει να τους στηρούμε. Ευχαριστώ, καλή τύχη. Λόγω στην κυρία Κρέζ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα για την, για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Συμφωνώ με κάποια τα σημεία που θέσατε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πετύχει αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαφθοράς και χαίρομαι με αυτό που είπατε, ότι ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι να χορηγηθούν πιο πολλοί πόροι για την καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος. Συμφωνώ, ωστόσο, και με κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκανε συνάδελφοί μου. Τονίζω ότι κάτι που λείπει, όπως είπε και ο κύριος Κάσμαν, ήταν ότι η ίδια λογική θα πρέπει να διέπει και το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Και θα ήθελα πραγματικά να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεσή σας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία. Ότι ο φόρος ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, δηλαδή ένας γενικός φόρος, δεν αποτελεί κάποια διάκριση κατά κάποιων συγκεκριμένων αγορών και ότι αποτρέπει την, ε, αν θέλετε, διακριτική μεταχείριση κατά κάποιων ε, αγορών. Κάτι άλλο, τα γενικό FTP θα βοηθούσε την εξαίρεση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το φόρο προστιθέμενη αξία. και τέλο θα ήθελα να κλείσω με το σχόλιο που έκανε και ο κύριος, ε, η κυρία Γερέρο ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε FTT σε παγκόσμιο επίπεδο ή μάλλον θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά θα έπρεπε πρώτα να, να ξεκινήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριος Σφέντσεν έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι κάπως έχω απογοητευτεί που δεν έχουμε μετάφραση από τα Σουηδικά προς άλλες γλώσσες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέβα για την έκθεσή του. 800 δισεκατομμύρια από τις αναπτυσσόμενες χώρες, το οκταπλάσιο από αυτό που χορηγούμε. Πώς τα δίνουμε τα χρήματα αυτά. Οι απαντήσεις νομίζω ότι τις δικαιούμαστε και μάλλον χρειάζεται βραβεία ο Νόμπελ. Αν μπορούμε να κατεβάσουμε στη γη το φεγγάρι, ας κάνουμε. Και τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Όσο υπάρχουν ηγέτες όπως ο Μουγκάμπε, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλους ηγέτες και άλλους δικτάτορες, αλλά εν περιπτώσει, το όνομα αυτό αρκεί για να σκεφτούμε. Γιατί ξέρουμε τι δυσκολίες είχε η Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες για να το σταματήσουν. Θα πρέπει, θεωρώ, να τονίσουμε πιο έντονα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί ιδάλω δεν τονίζουμε ποια είναι τα θεμέλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτές οι αρχές, αυτές οι αξίες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα όταν συζητάμε θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα δισεκατομμύρια αυτά που μετρούν, ξέρετε. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι αρχές. Ευχαριστώ κύριε Σβέντσον και τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Τζόνς, αν θέλετε σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ε, πιο έντονης προσπάθειας σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα να επενθυμίσω ε, κάποια μάλλον τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου, που τόνισαν τη σημασία και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη προτάσεις για μηχανισμούς καινοτομικής ε, χρηματοδότησης με δυναμικό προτέρων δημιουργίας ε, δυναμικού. Τα λαμβάνει λοιπόν αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά και την φορολόγηση του δυτικού τομέα, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανάπτυξη αναφέρεται ρητά σε θέματα φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα ως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πώς μπορεί να εφαρμόσει τέτοιους μηχανισμούς. Ευχαριστώ. Ο κ. Ε, Ντέβα έχει ξανά το λόγο, παρακαλώ. Έχω πολύ λίγο χρόνο, συγγνώμη. Δεν είδα ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή η Κομισιόν δεν είχε λάβει υπόψη αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι στις και δεν έχει πάει σε βάθος. Παρακαλώ λοιπόν να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη και προσπαθώντας να διατηρήσετε αυτά τα, τα λεφτά σε αυτέ τι αναπτυσσόμενες χώρε και σαν μηχανισμοί θα πραγματικά θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς οι οποίοι να εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα την εκλογή αυτών των χρημάτων. Όπως ο κ. Βάντσον είπε προηγουμένως, από πού έρχεται το χρήμα αυτό. Έρχονται από τις δικέ μα τράπεζε, από την Ευρώπη, έρχονται από το Λονδίνο, από το Λουξεμβούργο και πηγαίνουν αυτό σε παραδείσους φορολογικούς. Είναι λοιπόν, είναι χρήματα δικά μας είναι. Και βάζουν σε αυτούς τους παραδείσους αυτό το βρώμικο χρήμα, το οποίο χρήμα αυτό έρχεται από τις τράπεζές μας. Εάν πραγματικά πάτε στις τράπεζες μας και αν θέλετε να τις προστατεύσετε, όταν έγινε τρομοκρατία και η κρίση με την τρομοκρατία, εάν καταθέσετε πάνω από 5.000, λένε πού Πού τα βρίσκεται αυτά τα χρήματα πάνω από 5.000 ευρώ. Γιατί, γιατί κυνηγούσαμε αυτή, εκείνη τη στιγμή τους τρομοκράτες. Υπήρχε ένα κυνήγι των τρομοκρατών. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει, δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Υπάρχουν 500 δις που φεύγουν από μια ε, χώρα αφρικανική, 500 δις που φεύγουν, 50 δις που φεύγουν, ουδής ρωτάει τίποτα. Από πού έρχονται αυτά τα λεφτά κύριε Πρόεδρε της Αφρικανικής Αλφα χώρας. Εάν, εάν βάλουμε εμεί 5.000 ευρώ σε μια τράπεζα θα μας πούνε πού, τα βρήκατε αυτά τα λεφτά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μηχανισμός για την τρομοκρατία και αυτό ζητάω από την Κομισιόν να θέσει τον ίδιο μηχανισμό και για, τους, για αυτές τις χώρες που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να επανέλθω επίσης. Όσον αφορά τη φορολογία πρέπει να μπει επί των αγαθών. Για και έχω πει. Έχουμε το τσάι το οποίο, το οποίο εξάγεται. Ξέρετε αυτό το, το, το... Ξέρετε Ξέρετε από το τσάι που πληρώνεται από τα 2 ευρώ πόσα πέρα Μισό σέντς πηγαίνει στον παραγωγό. Μισό σέντς τα 199 και μισό που πάει. Δεν πάει στη Σρι Λάγκα. Κυκλοφορεί μεταξύ Λονδίνου και δεν ξέρω πού. Και θα πρέπει να δείτε πού κυκλοφορεί αυτό το χρώμα. Μισό σέντς πηγαίνει στη Σρι Λάγκα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πάνε σωστά στον κόσμο αυτό και θα πρέπει να διακρίνουμε να μην γίνουν τέτοιου είδου πράγματα. Και αν πραγματικά θέλετε να έχετε μια ε, καινοτόμο γνώμη και γνώση και άποψη από την Κομισιόν αυτό πρέπει να πράξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεβά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως προθεσμία κατάσταση των τροπολογιών είναι 19 Νοεμβρίου ενεστώτος στις 12 το μεσημέρι. Συνεπώς, ερχόμεθα στο επόμενο σημείο όσον αφορά την ανθρωπιστική η εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, η διάμεση ενασκόπηση του σχεδίου δράση και οι προοπτικέ. Θα ξεκινήσω εγώ την παρουσίαση με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, πρωτοβουλία, συγγνώμη, και αυτό αποτελεί συνέχεια μιας πρώτης που είχαμε, που είχαμε παρουσιάσει πριν λίγε εβδομάδε. Αν θυμάστε είχα παρουσιάσει εγώ μέσα σε αυτά τα πλαίσια τη ανθρωπιστική βοήθεια μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα επανέλθω σε αυτό που έχω πει. Όσον αφορά την εκπόνηση τη εκθέσεω. μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει η ανθρωπιστική ε, συμμετοχή τομή μη κυβερνητικών κυβερνήσεων κλπ. κλπ. η κυρία Τζόρτζεβα Κρυσταλίνα η οποία είναι επίτροπο και με τι. Ε, Υπηρεσίε Γενικής Διεύθυνσης 6. Όλοι αυτοί συμμετείχαν. Ε, το κόντεξ της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει επιβαρυνθεί, έχει χειροτερέψει και υπάρχει ε, ανάγκη μεγαλύτερης επέμβασης σε αυτό το θέμα το μέσο το οποίο, το εργαλείο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σχετικό και κρατάει αυτή τη στιγμή όλο το γόητρο το οποίο να έχει για τις επεμβάσεις αυτές. Το 2000 επίσης δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, επιστημιστική βοήθεια. Υπάρχει ένα φόρουμ για αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, καθώς επίσης το follow-up της συνένεσης καθώς επίσης ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ζητούν τη βοήθεια, πώς θα πηγαίνει αυτή και πώς θα περνάει μέσα από μια ασφάλεια αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όσον αφορά αυτό το μεγάλο πορτοφόλι, το σύνολο έχει διοργανωθεί και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός. Επιμένω όμως ότι κάθε ιδιαιτερότητα του κάθε εργαλείου θα πρέπει να παραμείνει ακέραιη Παραλλήλως βεβαίως να υπάρχει συνένεση και συντονισμός. Η συνθήκη της Λισαβόνα προβλέπει αυτό το πράγμα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία τη γενικης Διεύθυνση ΕΚΟ, εκο-οικολογίας δηλαδή, καθώς επίσης και οικονομίας και να μην μπερδεύεται αυτό το πράγμα με την πολιτική, εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΟΝ, καθώ επίση και τη Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τι μεγάλε κρίσει, μεγάλου ελληνικού κρίσει. Επίση θα πρέπει να δούμε πώ αυτή τη στιγμή η Κομισιόν μπορεί, όσον αφορά την έκθεση τη κυρία Ζανίκη, θα μπορούσε να δει κάτι παραπάνω και ότι αυτό το οποίο προτείνεται είναι αντίθετο από τα προτινόμενα στα πλαίσια της δική μας Επιτροπής και το γεγονός ότι αυτό να περάσει κινδυνεύει να πολιτικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια καθώς επίσης και μια μεταφορή, ε, μεταφορά συγγνώμη, των αρμοδιοτήτων της κυρία Τζόρτζεβα πράγμα το οποίο αντιταχθήκαμε πολλαπλώς εμείς. Ε, επίσης, Όσον αφορά στην συνένεση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για να ενισχυθεί η διαφάνεια του, η ορατότητα που υπάρχει σε όλα αυτά τα θέματα να εφαρμοστεί, καθώς επίσης και να πρέπει να υποστηρίξουμε, ώστε η συνένεση να γίνει αντιληπτή, να εφαρμοστεί, να είναι διαφανής και να γίνει γνωστή στο κοινό καθώς επίσης και ότι περιπλέκεται γύρω από αυτό. Επίσης, είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια δράση σε τομείς εκείνης οι οποίοι είναι ουσιώδη, ουσιώδη συγγνώμη, καθώς επίσης και να υπάρχει μια συνένεση για την εφαρμογή όλων εκείνων των συνετικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τα, ε, τις συστάσεις, τις οδηγίες κλπ. οι οποίες έχουν δει ε, αναφορά τη ανθρωπιστική βοήθεια, διότι είναι η ανθρωπική βοήθεια ανεξάρτητα οποιασδήποτε πολιτικής επέμβαση η οποία θα πρέπει να γίνει σε αυτά τα θέματα. Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει και την εφήρωή της καθώς επίσης και το βάρος της στο πολιτικό και το πολιτισμικό και θα πρέπει πάντοτε να προωθεί τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες. Η Κομισιόν και τα κάτι μέλη έχουν ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό να παίξουν όσον αφορά την υλοποίηση της των γενικών κατευθύνων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια ε, τις οργανώσεις. Καλό την Κομισιόν λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση όσον αφορά την προώθηση του ΔΕΙΑΣ, τη ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή, καθώς επίσης ε, παγόρευση οποιαδήποτε πολιτικοποίηση, ε, χρήση όπλων και ε, να πρέπει η βοήθεια αυτή να πηγαίνει όχι με τα προεφερθένα κριτήρια αλλά με βάση κατά πόσο οι χώρες αυτές είναι σε σημείο τέτοιο έφραυστο ή τροτό για να μπορούν να χρησιμοποιούνται για να μπορεί να υπάρχει ένα κοινό πεδίο εφαρμογής για όλες τις χώρες και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Επίσης μια εργασία η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, η οποία έχουν αλληλευθεί όσον αφορά τις ειδικού τομεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, για την Κομισιόν, για την προσπάθεια την οποία έχει πει και για του ομοφυλόφιλου επίση. Νομίζω ότι πραγματικά ότι αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα θέματος και εγώ επιμένω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ όσον αφορά την, την σεβασμό όλων εκείνων των παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και τι ανθρωπιδικέ προσπάθειε οι οποίε γίνονται σε διεθνέ επίπεδο και ενθαρρύνω περαιτέρω την, την εργασία η οποία επιτελούν αυτή τη στιγμή όλοι οι συμπράττοντε για να μπορέσουν καλύτερα να ενταχθούν μέσα σε αυτήν όλη τη διαδικασία θα πρέπει να θυμηθούμε όλε τι μεταρρυθμίσει που γίνανε στα πλαίσια του ΟΗΕ και το συντονιστή τη ανθρωπιστική βοήθειας η οποία έχει οριστεί για να υπάρξει μια προσέγγιση καλύτερη του κλάστερ καθώ επίση και τη συνεργασία με τι τοπικέ δομέ, τι πτυχές εκείνε κατατομή οι οποίοι υπάρχουν καθώ επίση και τη, συνεργασία, τη δυνατότητα συνεργασία μεταξύ κλάστερ Επίσης η, η δυνατότητα της διεθνούς συνεργασίας πέρα από την εψέψη στο σε αυτό το, θέμα. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής. Είναι ουσιώδες, οι δυνατότητες είναι να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται παρά κατ' εξαίρεση και μόνον σε ορισμένες πολίτικες περιπτώσεις. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια της ΕΕ καθώς επίσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ούτως ώστε ο σεβασμός και η εφαρμογή της, των οδηγιών του, του ΟΗΕ θα πρέπει να γίνονται απολύτως. Επίσης να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση ένθεν και κήθεν η προστασία ε, του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η πολιτική προστασία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να είναι συνεκτική, να υπάρχει συνένεση και να βοηθάει πάρα πολύ στην ανθρωπιστική βοήθεια την πραγματική την οποία δίδεται. Καλό λοιπόν την Κομισιό να παρουσιάσει προτάσεις νομοθετικού χαρακτήρα οι οποίες θα είναι φιλόδοξες για την πολιτική προστασία των χωρών αυτών καθώς επίσης και τη βελτιοποίηση όλων εκείνων των μέσων των οποίων υπάρχουν για τους πολίτες των χωρών αυτών και μια αμοιβαιότητα η οποία θα πρέπει να υπάρξει στα υπάρχοντα ήδη σχέδια. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την υιοθετία το Φεβράριο του 9 της νέας στρατηγικής η οποία υιοθετήθηκε όσον αφορά τη μείωση των καταστροφών σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά αυτές θα πρέπει αυτή θα πρέπει να τεθεί ε, σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν για να υπάρχει πιο συστηματική διάσταση όσον αφορά την πολιτική βοήθεια που δίνει σε αυτή τη χώρα καθώς επίσης και την ανθρωπιστική βοήθεια να υπάρχει ένας παραλληλισμός και μια συμπληρωματικότητα. Επιμένω πάρα πολύ επίσης ότι σε μικρή κλίμακα θα πρέπει να γίνει τη βοήθεια αυτή μέσα σε αυτά τα πλαίσια καθώς επίσης και να υπάρξει μια ε, οθέτηση, αν θέλετε όλων εκείνων των project τα οποία υπάρχουν μέχρι τούτε. Τέλος, λυπάμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ότι η πρόοδος η οποία έχει γίνει μεταξύ ανάπτυξης, αποκατάστασης και ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πάρα πολύ περιορισμένες μέχρι τούδε και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Επίσης η ευελιξία και η συμπληρωματικότητα δεν έχουν επαρκώς προχωρήσει. Θα ζητούσα λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και να υπάρχει επίσης και μια διασύνδεση και ένα, διασύνδεση συγγνώμη, και ένα, μια δυνατότητα μεταξύ του κατεπήγοντος και της ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία γίνεται όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, τα κράτη-μέλη και τις υπόλοιπες οργανώσεις. Δεδομένου η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ μικρή την οποία παρουσιάζω θα βρείτε αυτή τη στιγμή τροπολογίε, τροπολογίες οποίε έχω καταθέσει και τι έχετε αναχείρα στο φάκελό σας Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας, στα σχόλια και στις παρατηρήσεις σας, αλλά θα πρέπει να αναγγείλω πως η συζήτηση θα γίνει μετά την παρουσία της κυρίας Άστον, η κυρία Άστον η οποία είναι εδώ, άρα θα συνεχίσουμε μετά την ακρόαση που θα δώσουμε στην κυρία Άστον. Και περιμένω, ελπίζω, προσδοκώ τις δικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. J'en profite aussi pour laisser euh, με τις ευκαιρίες για να αφήσω, λίγο το, να αφήσω την Προεδρία στην Πρόεδρο η οποία έρχεται πίσω. Ευχαριστώ. Bonjour tout Γεια σας και πάλι όλοι. Έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να σα παρουσιάσω την κυρία Άστον, η οποία είναι αντιπρόεδρο τη Κομισιόν και η οποία είναι επιφορτισμένη για τι εξωτερικέ υποθέσει. Κυρία Άστον, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχή που βρήκα το χρόνο να έρθετε εδώ από τι επιτροπή μα για μια ανταλλαγή απόψεων. Η παρουσία εδώ ε, γίνεται μετά από την επίμονη δική μας ε, αίτηση να έρθετε εδώ αυτή τη στιγμή για να μας εξηγήσετε πραγματικά πώς ακριβώς γίνεται η συνεργασία για την ανάπτυξη μετά ιδιαίτερα την εισαγωγή της συνθήκης της Λισαβόνας καθώς επίσης και την υπηρεσία ε, η οποία δημιουργήθηκε για τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ. Ευχαριστώ. Ποτέ δεν τους αρκεί. En Όντως, ξέρετε αυτή η υπηρεσία εξωτερικών πράξεων, εξωτερικών δραστηριοτήτων θα γίνει υπεύθυνο όσον αφορά για την ανάπτυξη επίσης στην ΕΕ. Όλα θα μεταφερθούν σε αυτή ε, την την ειδική αρχή στην οποία εσείς προεδρεύετε και έχετε τη ευθύνη για την εξωτερική βοήθεια. Αυτή η μεταφορά λοιπόν μια ολόκληρης υπηρεσία στην εξωτερική δραστηριότητα όπως λέγεται τώρα αυτό μας οδηγεί στην απόφαση την οποία έχουμε λάβει για να δούμε πραγματικά τι θα γίνει με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και τη δημιουργία μιας καινούργιας Γενικής Διεύθυνσης. Είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή μας έχει πάρα πολλά ερωτήματα να σας θέσει. Γι' αυτό σπέβδω να σας δώσω το λόγο κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Συγγνώμη θα μιλήσω στα αγγλικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ε, στην Επιτροπή σας ότι ε, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας γιατί έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που εκλήθη να γίνω νότος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, πατή εκπρόσωπος και μέσα σε αυτή τη χρονιά έγιναν πολλά πράγματα. Ε, κυρίως όμως ε, εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε με τα διάφορα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα θέσουμε τα θεμέλια μιας Ευρωπαϊκής Πίεσης Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς και ιδιαίτερα σε εσάς κυρία Ζουτζολή, που πρόθυμα συνεργαστήκατε μαζί μου για να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαίρομαι που μπορώ, έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας το πώς βλέπουμε αυτή την υπηρεσία στο μέλλον. Αυτό που θα ήθελα καταρχήν να πω πάνω απ' όλα είναι ότι εγώ έχω αναλάβει την δέσμευση να εξασφαλίσω ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει στον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέει η συνθήκη και αυτό πιστεύω και εγώ για το μέλλον. Θα ήθελα σε μερικά λίγα λεπτά να σας πω ποιες θα είναι οι προκλήσεις για το μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε και πώς σκοπεύουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και μετά να δούμε και το πώς θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματική συνεργασία με τους υπόλοιπους επιτρόπους, ε, αλλά και με την Επιτροπή σας. Η εκρίζωση της ε, φτώχειας είναι ασφαλώς ο τελικός στόχος, όχι η μείωση της φτώχειας, η εξάλληψή της. Στόχοι Τη χιλιετίας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και ο Άντρε Πίμπαλξ όπως γνωρίζετε έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο από τότε που έγινε επίτροπος προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της χιλιετίας μαζί με τον πρόεδρο Μπαρόσο ε, ήταν παρόν στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου ο κύριος Μπαρόσο επανέλαβε την προσήλωσή μα στους στόχου τη χιλιετία. Θα πρέπει όμως ό,τι κάνουμε να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μέσα από ό,τι στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, μετά τη συνθήκη αβώνας είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε και να έχουμε την ανάπτυξη στο κέντρο της δράσης μας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δράσης, κάνοντας περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Ως αποτέλεσμα, έχουμε το εξής. Παλιότερα δεν είχαμε καταφέρει ε, να συνενώσουμε ε, τις διάφορες πτυχές της δράσης μας με τρόπο που θα μας επιτρέψει πλέον να κάνουμε Λισαβόνα. Αυτό δεν είναι επίκριση ε, προς οποιονδήποτε, προς οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Έτσι λειτουργούσαν τα προγραμματά μας παλιότερα. Σκεφτείτε τρία παραδείγματα. Πρώτον, αναπτυξιακό έργο στη Σομαλία. Ο κύριος Μπαρόσο προσπαθούσε να υποστηρίξει αυτή τη χώρα, να αποκτήσει ε, κυβέρνηση και να καταπολεμήσει την πειρατεία στα ανοιχτά των ακτών της. Από την άλλη μεριά, η IT, η δυνατότητα να κινητοποιήσουμε όλα τα κράτη-μέλη σε περίοδο κρίσης, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε ε, τις, τους που είχαμε, ε, μας βοήθησε να αντιδράσουμε γρηγορότερα. Όμως μπορούμε πολύ καλύτερα στο μέλλον, θα μπορέσουμε πολύ καλύτερα στο μέλλον. Τρίτο παράδειγμα, η Γάζα. Η ικανότητά μας να κινητοποιήσουμε ε, βοήθεια έτσι ώστε οι κάτοχοι, κάτοικοι της ε, Γάζας να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους και να ζουν από, αυτό, από αυτές τις εξαγωγές χρειάζονται χρειάζεται ε, τεράστιες προσπάθειες ε, σε μια περιοχή που το 85% ε, των κατοίκων ζουν χάρη στην ε, ε βοήθεια που αποστέλλεται και το 65% πληρώνεται από το κράτος. Συνεπώς είναι πολύ μεγάλο το έργο που έχουμε μπροστά μας στην εξάλληψη της φτώχειας και χρειάζεται να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας. ένα από τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ο Άντρισεν και εγώ να καθορίσουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Εγώ ως είπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν πρέπει να εξασφαλίσω ότι ο Επίτροπος Ανάπτυξης δεν θα έχει πλέον μόνο αρμοδιότητες για ένα κομμάτι του κόσμου αλλά για όλα. Για ό,τι κάνουμε στο πεδίο της ανάπτυξης. Γι' αυτόν τον λόγο ε, η απόφαση που πήρα η Κομισιόν το αναφέρει ρητά. Θέλουμε από κοινού με τον Άντρης να καθορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτη-μέλη, Κομισιόν, τα μέσα τα οποία διαθέτουμε και που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ό,τι είμαστε τώρα, χωρίς όμως, χωρίς, επαναλαμβάνω, να ε, παρεμποδίσουμε το έργο του Επιτρόπου Ανάπτυξης. Ε, ο Άντρης είναι πολύ καλός, θα τον υποστηρίξω και θα κάνει τη δουλειά του σωστά. Θα συνεργαστούμε μόνο εκεί που η συνεργασία μας θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και το γεγονός ότι εγώ είμαι και αντιπρόεδρος και είπατε εκπρόσωπος έχει σχέση με αυτό. Οι όσοι έχουν διαβάσει τη συνθήκη το έχουν καταλάβει. Ε, το θέμα αυτό περνάει και από μένα ακριβώς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Να κάνω και δύο άλλα εισαγωγικά σχόλια. Πρώτον, <clears throat> θα πρέπει να γίνουμε και πιο ευφυείς στη δράση μας. Συνεπώ πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά και με άλλες χώρες που ε, ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ε, Υπουργός Εξωτερικών κυρία Κλίντον το έχει πει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Όμως έχω συζητήσει τελευταία και με εκπροσώπους από την Βραζιλία και θα μπορούσαμε και με τη Βραζιλία να αναπτύξουμε τις, τη συνεργασία μας και με την Κίνα. Γιατί όχι. Τώρα, τελειώντα, θα ήθελα να αναφέρω τι τρει προκλήσει που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Πρώτον, εφαρμογή τη συνθήκη Λισαβόνα. Βρισκόμαστε στο τέλο τη πρώτη φάση, αλλά έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε πώ θα συνεργαστούμε, ιδιαίτερα στον τομέα τη ανάπτυξη και αυτό θα αποτελέσει τμήμα τη δράση μα για την εφαρμογή τη Λισαβόνα. Δεύτερον, πώ θα είμαστε όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Ε, ε, οι δικαιούχες χώρες ζητούν πιο γρήγορη αντίδραση από μέρους μας και πιο αποτελεσματική αντίδραση. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Το ακούω, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το κατά πόσον μερικές χώρες είναι πιο γρήγορες από την μια μεριά αλλά χωρίς να είναι πλήρεις και αποτελεσματικές στην βοήθειά τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τρίτον, τρίτη πρόκληση η ευελιξία. Γιατί, Γιατί ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, ταχύτατα και χώρες και θέματα που δεν ήταν στην ατζέντα μας πριν από μερικούς μήνες ξαφνικά γίνονται, μπαίνουν στην ατζέντα μας. Η Εμένη για παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το θέμα της ασφάλειας μας ε, ε, ανέδειξε το θέμα της Ιεμένης. Η, Ιεμένη ε, έχει πολλά προβλήματα φτώχειας. Είναι μία από τις χώρες που θα μπορούσε να μείνει άνυδρη τα επόμενα χρόνια. Έχουν με πολλά προβλήματα διαλόγου αυτή τη στιγμή με την Ιεμένη κλπ. Συνεπώς, η φτώχεια και η ανέχεια επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλούς δρόμους, από πολλούς δρόμους και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους. Μία από τις προκλήσεις μας λοιπόν θα είναι να δούμε πώς θα εντάξουμε στο σύστημά μας την ευελιξία και πώς θα κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι ώστε να βλέπουμε πέρα από τι χώρε που είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σε χώρε που ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν πρόβλημα στο μέλλον, σε χώρε όπου υπάρχουν θύλακες φτώχειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά ω εισαγωγικά σχόλια προς Ανατολισμό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σα. Θα ήθελα να έχω έρθει πιο νωρί. Ε, δυστυχώς η ατζέντα μου δεν το επέτρεψε. Όμω, η καθυστέρηση αυτή δεν σημαίνει ότι βάζω σε δεύτερη γραμμή τα θέματα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Lady Ashton. Ευχαριστώ, Lady Ashton. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους κάνους του παιχνιδιού. Για να γίνει μια πραγματική συζήτηση, ένα πραγματικός διάλογος, ε, θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Θα ήθελα να, πα... να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας στο 1,5 λεπτό, λεπτό συνάδελφοι. Ε, θα... Έχουμε ομάδες τριών ε, συναδέλφων ε, που θα μιλούν και θα δίνω μετά τον ε, λόγο στην κυρία Στυλέδη Άστον για να απαντήσει, όχι περισσότερο από 8 λεπτά όμως. Ο λόγος καταγίνει στην κυρία Στρίφλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ, κυρία, Πρόεδρε, κυρία Άστον. Τα ανθρωπιστικά, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτή τη στιγμή το πιο βασικό πράγμα που μπορεί να κάνει η ΕΕ σαν αυτέ τι φυσικέ καταστροφέ οι οποίε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αυτή τη στιγμή μια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να για τι εξωτερικέ υπηρεσίε για να υποστηρίξει τη Γενική Διεύθυνση τη Οικολογία και να μην υπάρξει μια πολιτική εκμετάλλευση αυτού του θέματος, Πακιστάν, ε, Αϊτή κλπ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η διαστρωτική παρέμβαση μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τόσο, αλλά και η συνένεση που είχε βρεθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται στην εσχάτη, περισσότερο έσχατο καταφύγιο εφόσον υπάρχει ανάγκη σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστροφών και ζητήθηκε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ της δικής υπηρεσίας καθώς επίσης και της υπηρεσίας, των υπηρεσιών της Κομισιόν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κυρία Ντεκάιζερ έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε κυρία Άστον. Ευχαριστώ που είστε εδώ κυρία Άστον. Η ερωτήση μου έχει σχέση με τη συνεργασία που έχουμε με τον ΟΗΕ για την παρατήρηση των εκλογών, παρακολούθηση των εκλογών, συγγνώμη, ιδιαίτερα όσον αφορά το Σουδάν. Εάν για τις εκλογές που γίνονται στο Σουδάν τον Απρίλιο ενεστώτος είχαμε ορισμένες δυσκολίες στην αρχή με τις σχέσεις τις οποίες αναπτύξαμε με τον ΟΗΕ ιδιαίτερα όσον αφορά την κάλυψη υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ και τη δυνατότητα των τη δυνατότητα των παρατηρητών μας να πάνε στα νοσοκομεία του ΟΗΕ και σε άλλους χώρους του ΟΗΕ και η δυνατότητα εκένωση από αυτή τη χώρα εν χρειαστεί έγινε μία κοινή συνεννόηση και μία συνένεση μεταξύ ΟΗΕ και ΕΕ. Το να γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύετε από τότε οι σχέσεις μας με την ΟΗΕ έχουν διευκρινιστεί και κατά πόσον εμείς σαν παρατηρητές έχουμε την πλήρη συνεργασία με τον, με τον ΟΗΕ γιατί είναι θέμα ασφαλεία για την επόμενη αποστολή που θα σταλεί στο Σουδάν. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκέρεντς έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ όσον αφορά την καλή ανάπτυξη, σωστή ανάπτυξη για το, το θεσμική ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να σου το πω εξ και διαζώσεις. Η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει πολύ ευγενείς και πολύ συγκεκριμένους στόχους. Έχει στόχους και δεν είναι μόνο τα μέσα, αλλά έχει και στόχους και υπάρχουν, ε, υπάρχουν καταστάσεις ότι πραγματικά δημιουργείται μια σύγκρουση γιατί ο πόλος ανάπτυξης ε, σε αυτό τον πόλο αντιτίθεται μια άλλη αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς αυτή η διαμάχη η οποία δημιουργείται μεταξύ των διαφόρων φορέων θα λυθεί, θα επιληθεί. Και δεύτερη ερώτηση, μήπως δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση ούτω ώστε να κάνουμε ένα κατάλογο αυτών των συγκρούσεων των συμφερόντων και εντό με 6, 9 ή 12 μηνών να βρούμε έναν επίτροπο, τον Επίτροπο Αναπτύξεως, Ανάπτυξη παραδείγμα, πώς μπορεί να μας πει Κατά πόσο, εφόσον συνεχιστούν αυτές οι συγκρούσεις που υπάρχουν, δεν εμποδίζεται το έργο το οποίο επιτελεί, πώς μπορεί να είναι διαφανή όλα αυτά, καθώς επίσης και μια διαχείριση όλων αυτών των συγκρούσεων. Και να συζητεί εδώ ένα από τι επιτροπές μου. Επίση, ανησυχώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ότι εξασθενεί όλο και περισσότερο το Συμβούλιο το οποίο όσον αφορά το θέμα της πολιτικής και την ανάπτυξη έχει ένα ρόλο να παίξει καθότι πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος είναι κατά το ίμιση δικό του και κατά το ίμιση άλλων και διαρωτώτε κανείς κατά πόσον εσείς προσωπικά μπορείτε να μας πείτε ότι δεν έχουμε άλλον ε, συνομιλητή και ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εσείς θα μας το πείτε αυτό το πράγμα ε, το Συμβούλιο θα μπορούσε να είναι παρόν σε τέτοιου είδου συναντήσει, ούτω ώστε να δίνει την άποψή του, διότι δυστυχώ δεν είναι παρόν. Και λέει, Άστον έχει το λόγο, παρακαλώ. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τι ερωτήσει για την κυρία Τρέιφλερ. Για μία γενική διεύθυνση ΕΚΟ για την ε, Υπηρεσία Πολιτική Προστασία. Είναι σημαντικό φυσικά η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να μπορεί να λειτουργήσει πέρα από κάθε συνάρτηση με οτιδήποτε στρατιωτικό θεωρώ ότι θα πρέπει να καθορίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λειτουργήσουμε. Είδαμε στην ΑΕΤ ότι η δυνατότητα των κρατών μελών να παρέχουν ε, πλοία, ε, παραπήγματα για νοσοκομεία, να παρέχουν δυνατότητα προσγείωσης ε, του εξοπλισμού χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στο έδαφος ήταν απαραίτητα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να κινητοποιηθούν με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης. Το ερώτημα λοιπόν που πάντα θα ανακύπτει και θα είναι και μάλιστα δύσκολο πάντα και σημαντικό σε οποιαδήποτε καταστροφή είναι το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα έχουμε στη διάθεσή μας με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και με την συνάδελφο συνεργαζόμαστε με την κυρία Γεωργίευα συνεργαζόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε η μία να υποστηρίξει την, άλλη για την άμεση ανταπόκριση σε ό,τι αφορά τα θέματα συντονισμού για το Πακιστάν, για παράδειγμα, όπου τα κράτη-μέλη και οι πόροι του Συμβουλίου, οι πόροι της Επιτροπής πρέπει να συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς πρέπει να πετύχουμε και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφής για το ποιος είναι ο ρόλος και η αρμοδιότητα καθενός. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ο συντονισμός αυτός. Εν μέρη, όπως έγινε στο Πακιστάν και στην ΑΕΤ. Και εν μέρη, ορίζοντας ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για το μέλλον. Και κοιτάμε λοιπόν πώς μπορούμε στο Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουμε για τον καλύτερο σκοπό με την καλύτερη αποτέλεσμα τους πόρους αυτούς. Κυρία Ντεκάιζερ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το έργο σας και σας ευχαριστώ που συμφωνήσατε να ηγηθείτε των προσπαθειών και πάλι. Για να αναφερθώ στα τελευταία σας σχόλια. Σύμφωνοι, δεν μπορούμε να δράσουμε χωρίς το τμήμα της ασφάλειας. Μίλησα με τον πρόεδρο Μπέκη χτες για τις δραστηριότητές του. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα, γιατί η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Κυρία Γκέρεντς, για τους ευγενείς σκοπούς συμφωνώ. Συμφωνώ και για την επίτευξη των στόχων. Δεν θέλω να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και της ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα της ε, υπηρεσίας. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ υπό ποιε συνθήκε θα βρισκόμασταν σε σύγκρουση και όχι επειδή είμαι αφέλη. αλλά γιατί πολύ απλά δεν θεωρώ ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τη συνθήκη τη Λισαβόνα εάν βρεθούμε να έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό που συμβαίνει ήδη είναι ότι ο άντρα και εγώ συζητάμε κάποια θέματα και κοιτάμε πώ μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουμε του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα και πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους ανάπτυξης σε συνάρτηση με τα άλλα εργαλεία. Ένα καλό παράδειγμα για τις δραστηριότητες κατά της πειρατείας στη Σομαλία. Η υποστήριξη των χωρών που έχουν πληχθεί λόγω της πειρατείας, η υποστήριξη της Σομαλίας όπου μπορούμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια με διάφορες όμως δράσεις. Αυτό που κάνουμε δεν είναι απογραφή εγώ και ο κύριος Πίγκμπαλξ ε, καταρτίζουμε το πρόγραμμα και θα πρέπει να συνεργαστούμε για τους στρατηγικούς στόχους, αλλά και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Να υπάρχει μια συνέργεια των μέσων όπου είναι αυτό δυνατόν. Και χαίρομαι που ενδιαφέρει αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ίσως να υπάρξουν τέτοιοι τομεί σύγκρουσης. Δεν το πιστεύω, αλλά αν διακρίνουμε τέτοιους τομείς, εγώ και ο κύριος Πίμπαλξ θα το λύσουμε το θέμα αυτό, γιατί χωρίς αυτή την συνέργεια όλοι αυτοί οι ευγενείς στόχοι που αναφέρετε δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία voorzitter. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω τις ερωτήσεις του κυρίου Γκέρενς για την αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία αποτελεί έναν πολιτικό κλάδο του αθλήματος. Γι' αυτό λοιπόν και αγωνιζόμαστε εδώ πέρα για το ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό της επίσημης αθλητικής βοήθειας ε, και του EDF. Είπατε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σύντομα τέτοια σύγκριση. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από τις ε, εταιρικές σχέσεις τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνοχή του άρθρου 208 αν βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές οι αντιπροσωπείες πρέπει να επιδιώκουν εμπορικούς στόχους και την προηγούμενη φορά που καλέσαμε τον Βέλγο Υπουργό Αναπτυξιακής Βοήθειας δεν ήρθε γιατί είπε ότι δεν είμαι εγώ πλέον αρμόδιος η Λέτη Άστον είναι πλέον αρμόδια και επειδή είναι τόσο πολιτικό θέμα η αναπτυξή η αναπτυξική βοήθεια είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι πλέον δεν έρχεται Υπουργό Αναπτυξιακή Βοήθεια και η Λέδη Άστον δεν έρχεται γιατί δεν έχει χρόνο. Πώ θα το λύσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και πώ ε, θα μα ε, δείξετε το σεβασμό που μα αρμόζει και εσεί αλλά και ο αντίστοιχο και αρμόδιο Υπουργό του Βελγίου. Ευχαριστώ. κύριε κύριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Lady Ashton Κάθη. Έθεσε ένα ερώτημα. Ρώτησε κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα τα θέματα αναπτυξιακή βοήθεια με πιο καλή διακυβέρνηση, ευελιξία. Να απαντήσω ότι ναι, θεωρώ ότι κάποια από τα συστήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρχαϊκά, γιατί είχαν δημιουργηθεί και είχαν ε, ξεκινήσει την δεκαετία του 80 δεν διέπονται από τις σύγχρονες ε, διατάξεις διαφάνειας, ε, ευελιξίας κτλ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν αν αλλάξουμε κάποια από τα συστήματα που επικρατούν. Σήμερα στον εταιρικό τομέα και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ λοιπόν σε ό,τι αφορά την καινοτομική χρηματοδότηση. Μήπως είναι μια μεγάλη πατάτα, γιατί δεν έχουμε τέτοια εκατοντάδες δισεκατομμύρια να δώσουμε στον κόσμο Χρειαζόμαστε όμως πιο πολλά χρήματα. Όπως ξέρετε η Βρετανική κυβέρνηση συμφώνησε για το αλλά ξέρετε, για το 0,7% αλλά από ό,τι ξέρετε αυτό δεν αρκεί. 800 δισεκατομμύρια λοιπόν ευρώ φεύγουν παράνομα προς φορολογικούς παραδείσους από τις αναπτυσσόμενες χώρες και εμείς σε αντάλλαγμα τους δίνουμε 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακή βοήθεια. Αν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά έμεναν στις αναπτυσσόμενες χώρες, αν αυτά τα 800 δισεκατομμύρια ε, χρησιμοποιούνταν για την εξάλληψη της φτώχειας, για τις εμπορικές πρακτικές, για τα ε, δικαιώματα τα τετρικά στις χώρες αυτές, θα σημειώναμε τεράστια πρόοδο. Ας συνεργαστούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ, έχετε λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ζητήσω συγγνώμη που ξαράργησα. Το αεροπλάνο μου προσγειώθηκε πριν από μία ώρα μόλις. Να πω προς την ε, ύπατη εκπρόσωπο ότι είμαι εισηγητή για την ε, προτινόμενη ε, αναθεώρηση του DCI. Και ήμουν και υπεύθυνο και για την ενδιάμεση αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τους φόρους για το θέμα αυτό. Το, το Κοινοβούλιο ψήφισε τη σχετική νομοθεσία και τώρα πια δεν συζητάμε Δεν, λέμε, δεν μιλάμε πλέον για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Βρισκόμαστε στη φάση μετά τη Λισαβόνα και εγώ ξέρετε δύο φορές ε, ε, περιπλανήθηκα στο Δουβλίνο και μίλησα στον κόσμο για την συναπόφαση. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να δώσει τις αρμοδιέ του σε, την, ε, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η υπηρεσία εξωτερική δράση εσείς θα υποβάλλετε κάποιες εφαρμόσιμες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε κύκλους. Και ξέρετε, είμαστε πλέον φορέας με συναπόφαση στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος και πάλι στη ε, Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Σαρτζεντίνη, ε, δεν απάντησα προηγουμένως στη δεύτερη στο τμήμα του κύριου, κύριου του και τώρα με ευκαιρία το δικό σχολείο θα το κάνω. Εγώ ήμουν παρούσα στην ε, έκτακτη συνεδρίαση στο άτυπο στο Συμβουλίο των Υπουργών ε, ανάπτυξης και πλέον η ε, οι Υπουργοί Ανάπτυξης πρότεινα να συναντιόνται μισή μέρα μόνοι τους ε, επισήμως και όχι μόνο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. δεν έγινε πολύ γνωστή αυτή η πρόταση, αλλά είναι αλήθεια και μάλιστα είναι δεκτή και ε, ήδη προγραμματίσαμε ε, μια τέτοια συνάντηση στο πρώτο μισό της Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει τα κράτη-μέλη να δίνουν την άποψή τους και ε, πρέπει τα κράτη-μέλη να μιλάνε σε μένα, να μιλάνε στην Κομισιόν, να μιλάνε σε εσά. Και να υπάρχει ένας, ένα νήμα που θα συνδέει όλες αυτές τις δράσεις. Και έτσι θα εξασφαλίζουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο κ. Μισελ, ε, αρνήθηκε να έρθει εδώ να σας μιλήσει, παρόλο θα το ήθελε, ακριβώς διότι ακόμα δεν έχουμε ε, βελτιστοποιήσει το σύστημα διαλόγου και συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το κάνουμε. Ο Άντρης πάντοτε είναι παρόν στα Συμβούλια Υπουργών ανάπτυξη. Η κυρία Ζολή ε, παρούσα στο άτυπο Συμβούλιο. Ο κύριος Μισελ επίσης ε, θα είναι. Ε, συνεπώς στο μέλλον θα λάβει το όλο σύστημα μια πιο σαφή μορφή. Ε, νομίζω ότι θα βρούμε μία λύση στο μέλλον. Τώρα, ε, ε, για τη διαφάνεια. Πράγματι, το είναι πολύ σημαντικό να δούμε το πώς θα εξυγχρονίσουμε τη δράση μας, πώς θα την κάνουμε πιο ευφύ. Και θα πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές, οτιδήποτε έχει, κάποιοι έχουν κάνει διαφορετικά. Εγώ στο παρελθόν μου Έχω πάρει παράδειγμα από το πώς οι επιχειρήσεις ε, έχουν χειριστεί θέματα ε, ανάπτυξη δραστηριοτήτων και modeling και ε, δημιουργίας μοντέλων. Νομίζω ότι έχει ξεκυλήσει επί, Μισελ ή ο διάλογος. είναι πολύ σημαντικό όμως στο πλαίσιο της διαφάνειας να εξασφαλίσουμε και καλή διακυβέρνηση. Γιατί μέσω καλής διακυβέρνησης μπορούν να ρυθμιστούν πολλά θέματα διαφάνειας. Ταυτόχρονα έχω ήδη ξεκινήσει να σκέφτομαι τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση και σίγουρα θα το δείτε και εσείς και θα το δούμε και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη αυτό το θέμα θα, ο κ. Πίμπαλξ θα τεθεί επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Για το θέμα των πράξεων κατεξιοδότηση, ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσπαθούμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση. Εργάζομαι σκληρά σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους αρχή πίσω από, το, βασικό θέμα πίσω από όλα αυτά τα νομικιστικά ζητήματα είναι πώς θα συνεχίσουμε να α, συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο, πώς θα συνεχίσει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαδικασία προβληματισμού. Εκεί όμως που δεν εξασφαλίζω συμφωνία πρέπει να βρω μια ρεαλιστική λύση. Και γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν μπλοκαριστεί έτσι και πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Θα προσπαθήσουμε. Από τη συνάντηση του Στρασβούργου φάνηκε ότι υπάρχει διάθεση να βρούμε μια έξυπνη λύση έτσι ώστε και το Κοινοβούλιο να έχει αυτά που χρειάζεται χωρίς να ε, μπλέξουμε με τους ε, δικηγόρους και με νομικά επιχειρήματα. Ευχαριστώ κ. Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λέτε Άστον, ε, δύο ερωτήσεις. είχα παρουσιάσει αυτή τη στιγμή και θα το προσθέσω και σήμερα για την Αιθιοπία, την τελική κρίση που έπρεπε να κάνουμε εκεί. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο για τη θέση όσον αφορά το μέλλον της, ε, των, απο, των αντιπροσωπιών που στέλνουμε εκεί, των αποστολών που στέλνουμε εκεί, πώς θα το χρησιμοποιήσετε αυτό έτσι όπω είναι, θα είναι αμερόληπτη, ανεξάρτητη, για τη διαδικασία εκλογών που γίνεται εκεί και θα ακολουθούν τις δικές μας οδηγίες και θα έχουν σαν σκοπό να προστατεύσουν τα βασικά δικαιώματα των πολιτών εκλέγοντας ελεύθερα τους ηγέτες τους. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για το ρόλο αυτών των εργαλείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την παρατήρηση, παρακολούθησε και την αρχιτεκτονική κατά πόσον η Κομισιόν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία δεν γίνανε πολύ καλά και ανήκουν σε δύο χώρους διαφορετικώς. Όσον αφορά τη βοήθεια για την επίσημη βοήθεια για την ανάπτυξη, ξέρετε, λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε λόγω δίδεται βεβαίως λόγω, ε, σαν ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό είναι ένα πλήγμα και ένα άλλο πλήγμα από κρατημέλη έρχεται το οποίο με πολλά κράτη θέλουν αυτή τη στιγμή να βάλουν ε, ε, μέσα στη βοήθεια αυτή είναι την διατήρηση της ειρήνης, τη διαφύλαξη ειρήνης και τώρα εφόσον ετοιμάζουμε τον, τον προπολογισμό του 2011 βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το βασικό θέμα δεν είναι η ανάπτυξη, δεν είναι βοήθεια, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο το οποίο επισέρχεται. Ποια είναι η θέση σας αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να προστατεύσετε αυτή καθε αυτή τη βοήθεια η οποία γίνεται για την ανάπτυξη και μόνο και όχι άλλους λόγους. Ο κ. Κάσμαν έχει παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε είναι πάρα πολύ ευτυχής που σας βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Ένα σχόλιο το οποίο είπα προηγουμένως όσον αφορά τις εξωτερικές αποστολές της παρακολούθησης. Εγώ θα πρέπει να πω ότι υπάρχει αυτή η αντιπροσωπεία που είναι πάρα πολύ μικρή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι αυτό δεν είναι κατά να προστατεύσει τις αρχές οι οποίες έχουν. Πώς η Επιτροπή εν αυτή εδώ έχει πει ότι θα πρέπει να περικοπούν και το άρθρο 8 λέει αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδιαίτερα να αφορά τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Βλέπω λοιπόν ότι σε πολλές χώρες ε, εξωτερικές αλλά και συνέψε αυτά τα πράγματα θυσιάζονται τα οποία σας ανέφερε. Έτσι λοιπόν στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έρχεται ένα κείμενο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέξεις όσον αφορά τους ομοφιλόφουλους γιατί υπάρχουν μορφωτικές πολιτιστικές διαφορό. Πώς πραγματικά μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μια εξαίρεση όσον αφορά την παγκοσμιότητα των ανθρωπίων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα για στην ΕΕ και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξαιρέσουμε στα 27 μας στις 27 μας χώρες αυτό το πράγμα. Αυτό που με ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι ότι ενώ το Κοινοβούλιο έχει πει αυτή τη στιγμή έχει πει ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια εξαίρεση και θα περιλαμβάνει το οπωσδήποτε το δικαίωμα των ομοφιλοφίλων μέσα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ μια ερώτηση. Εγώ είχα δεχθεί τον προσωπάρχη σα που έδειχνε πραγματικά ποια δομή θα έχει αυτή η εξωτερική αποστολή. Σε αυτό το οργανόγραμμα υπάρχει μία οργάνωση με τέσσερα θεματικά, θεματικές υπηρεσίες τύπματα. Διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη δεν υπάρχει σε αυτό το οργανόγραμμα, καθώς επίσης και η απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία δίνει σε εσά την δυνατότητα για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη. Σημειώνω ακόμη, οι χώρες ΑΚΕ, οι οποίες δέχονται πολύ περισσότερο από το μισό από αυτή τη συνεργασία δεν υπάρχει καν μέσα. Επίσης η ομάδα εργασίας του Κοντεύ και, ε, και δεν υπάρχει μέσα στη δομή στο οργανόγραμμα αυτό. Έτσι λοιπόν αυτή η πολύπλευρη θυματική κατάτμιση η οποία γίνεται στο οργανόγραμμα ε, θα πρέπει να συλλαμβάνει τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις καθώς επίσης και την ισότητα των δύο φύλων. Εν ταυτό βεβαίως την προγραμματισμό τη Γενική Διεύθυνση της Ανάπτυξης γίνεται μια, μια μεταφορά από αυτήν προ τι εξωτερικέ υποθέσεις προς τις εξωτερικές υποθέσεις πράγμα το οποίο χάνει τη δυνατότητα που είχε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Κατά πόσον αυτό αληθεύει κυρία Άστον ότι έτσι είναι τα πράγματα και κατά πόσον εσείς θέλετε να διατηρήσετε την, την πραγματογνωμοσύνη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανάπτυξη, πράγμα το οποίο έχει γίνει διακτό από τη διεθνή κοινότητα και θα πρέπει να συνεχιστεί όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και πώς εσείς θα, θα εγγυηθείτε ότι όλα αυτά τα οποία προβλέπω στη Συμφωνία της Λισαβόνος θα γίνουν σεβαστά και θα ε, εφαρμοστούν. Ε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. <laughs> thank you very much again. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Εμπερμαν. Ξέρω ότι είναι η έκθεση σας σήμερα και δεν έχω ακόμα δει τι έχει γίνει. Αλλά είμαι βέβαιη ότι θα ήταν μεγάλη επιτυχία και δυστυχώς ε, δεν είσαστε σε θέση να υποβάλλετε την τελική σας έκθεση. Αυτό που είπατε και το οποίο έθιξε και ο Μάικλ για τις ε, ε, αποστολές παρατηρήσεις εκλογών. Το έθιξε και η Βερονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα και η θέση αυτή ακόμα δεν έχει δημορφωθεί όπως θα ήθελα. Καταρχάς πρόκειται για ένα θεμελιώδες ε, στοιχείο και μια θεμελιώδης πτυχή των όσων κάνουμε. Καταδεικνύεται έτσι η δέσμευσή μας στην πραγματική δημοκρατία και θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε κατά πόσο ήταν δίκαιες ή μη οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αποτελεί ένα βασικό μήνυμα που αποστέλουμε προς τον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει αυτά που λέει. Θέλω λοιπόν να αναπτυχθεί περαιτέρω το στοιχείο αυτό. Δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να το σκεφτώ όσο θα έπρεπε. Γιατί ήθελα πρώτα να μιλήσω και με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που έχουν πάει ως παρατηρητές και ξέρουν τι συμβαίνει επί τόπου, όπως και εσείς ξέρετε τι σημαίνει να αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Και να κοιτάξω πιο προσεκτικά το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι σωστοί πόροι για το σωστό σημείο. είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει στο Σουδάν και είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση ασφαλώς. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε δεν έχω έξυπνες ευθύς απαντήσεις, αλλά ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε να τις καταρτήσω. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η πτυχή αυτή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα, για αυτά που είπατε για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και θεωρείτε ε, ότι αν θέλετε, στηβάζονται τα προβλήματα. Έχετε φυσικά δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σαφείς για αυτά που κάνουμε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, η συνεργασία με τι βιομηχανοποιημένε χώρε. Όλα αυτά είναι σημαντικά και για τι αναπτυσσόμενε χώρε, οι οποίε χρήζουν βοήθεια και χρειάζονται του πόρου μα. Και το εύρο του τι σημαίνει βοήθεια αναπτυξιακή, από το να βοηθήσουμε τον κόσμο να ζήσει, μέχρι το να δοθούν οι ευκαιρίες για την σωστή αξιοποίηση των πόρων με βιώσιμο τρόπο θα αποτελέσει μία άλλο ένα και πιο μεγάλη πρόκληση για το μέλλον και θα πρέπει να είμαστε σαφείς και να ξέρουμε τι πρόβλημα ε, αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και πώς θα το επιλύσουμε. Μάικλ, αναφέρθηκα στα πρώτα ερωτήματα που έθεσες. Ξέρετε ποιες είναι οι θέσεις μου για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τι θεωρώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι κανείς ε, άνθρωπος και να είναι εδώ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο, δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφοροποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σαφεί και ε, άκαμπτοι σε αυτά που πιστεύουμε. Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι θέματα που μας απασχολούν, όπως θέματα φύλου, εθνότητας και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται να θεωρήσουμε ότι κάποια θέματα είναι πιο σημαντικά από άλλα. Πρόκειται για μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε σε κάποια τμήματα του κόσμου. Το ξέρετε αυτό. Είναι μια πρόκληση την οποία προσπαθούμε να θέσουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Και αυτά μπλέκονται, ξέρετε, και με άλλα θέματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξακολουθώ να έχω την διάθεση και την δέσμευση να δραστηριοποιηθώ γι' αυτό. Καταλαβαίνω λοιπόν τι ανησυχίε σα, κυρία Ζολή, τώρα θίξατε πολλά θέματα. Να προσπαθήσω να εξηγήσω το εξή. Θα υπάρξει μια γενική διεύθυνση DEFCO η οποία θα, θα δημιουργηθεί. Δεν πρόκειται να ξεφορτωθούμε λοιπόν το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να χαθεί στο οργανόγραμμα, το ενδεικτικό οργανόγραμμα. Γι' αυτό άλλωστε είναι και ενδεικτικό οργανόγραμμα. Ήταν μια πρώτη απόπειρα να περιγράψουμε την κατάσταση, αλλά μόνο εν μέρη δεν περιγράφεται, για παράδειγμα, πλήρως το γεγονός ότι η εκπεριτροπή Προεδρία εξακολουθεί να ηγείται τη ομάδα εργασίας ε, για την ανάπτυξη. Γι' αυτό δεν είμαστε παρόντε, γιατί υπάρχει αυτή η εκπεριτροπή Προεδρία. Δεν έχουμε ξεχάσει λοιπόν τα θέματα αυτά, πολύ απλά όμω δεν περιλαμβάνονται στο EAS. Προσπαθούμε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ να βρούμε ποιες θα είναι οι αντιπροσωπείες ε, στην υπηρεσία εξωτερική δράσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να δούμε και ποιο χρονοδιάγραμμα θέλουμε να ακολουθήσουμε. Θέλουμε ο κόσμος να μάθει πιο πολλά σχετικά με το τι κάνουν αντιπροσωπείες μας σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να συμπεριληφθούν και αυτοί. Και η τεχνογνωσία μας φυσικά. Θα δείτε λοιπόν ότι η εμπειρογνωμοσύνη θα παραμείνει στην ΤΕΦΚΟ, θα υπάρχουν γεωγραφικά γραφεία στο EAS, θα συνδυαστούν οι προσπάθειες και θα είναι σαφέ το ποια είναι η αρμοδιότητα του άντρε της Κρυσταλίνα. Το οργανόγραμμα όμω που καταρτήσαμε περιγράφει μόνο ένα τμήμα της όλης ε, κατάστασης και μόνο στο τέλος θα προκύψει ένα άθροισμα των επιμέρους μερών. Δεν προσπαθούμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τον σαφή και ξεκάθαρο ρόλο του Επιτρόπου ως αντιπρόεδρος, ως πρώτη αντιπρόεδρος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το τονίσω αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύνδεση προκειμένου οι αντιπροσωπείες, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να μπορούν να συνεργαστούν με τον άλλο τρόπο. La parole est maintenant à Monsieur Vergel. Hvala θα ξεκινήσω λέγοντας ότι με χαρά μου βλέπω ότι η Λέδη Άστον είναι όλο και πιο χαλαρή στο ρόλο της. Κάθε φορά που τη βλέπω, τη βλέπω όλο και πιο άνετη. Τα αναπτυξιακά ζητήματα σίγουρα συνδέονται στενά με πολιτικά θέματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σαφή πολιτική θέση εκεί που αυτά τα δύο, το πολιτικό με το αναπτυξιακό, αλλά επικαλύπτονται. Υπάρχουν θέματα, μεταξύ των οποίων ορισμένα τα οποία αναφέραμε σήμερα, που χρειάζονται άμεση απόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να λύσουμε πολιτικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Για παράδειγμα, Δυτική Σαχάρα πολύ επικαιρό ζήτημα. Αύριο θα έρθει στην επικαιρότητα το Κασμίρ. Η Εμένη είναι επίση θερμό σημείο του πλανήτη. Όχι, γιατί όχι εξαιτία αυτών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή για πολύ καιρό οι ε, κάτοικοι τη Εμένη ε, βομβαρδίζονται. Ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει γίνει ρουτίνα. Επίση, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Γάζα, Γάζα. Ε, χαίρομαι που αναφέρετε τη Γάζα πάντοτε στις ομιλίες σας. Νομίζω ότι το μέσο των ειδικών αντιπροσώπων που έχει γίνει πλέον ρουτίνα είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει να βρούμε πιο αποτελεσματικά μέσα. Ευχαριστώ. Merci, Madame Grèce. Ευχαριστώ, Κύριε Ευχαριστώ την κυρία Σνούμ Ευχαριστώ που είστε εδώ αυτή τη στιγμή. Η εξωτερική υπηρεσία δεν έχει μια συνοχή όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν άπτονται πολλών τομέων, γεωργίας, αλληλείας κλπ. Θα ήθελα να παραφέρω όμως στη βιοπειρατεία. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια λαιλάτιση όλων εκείνων των φυτών τα οποία αρπάζονται από αυτές τις χώρες, τα οποία χρησιμοποιούνται για αισθητικούς, καλλιστικούς και άλλους λόγους, σαν καλλιτικά. Πρόκειται λοιπόν εδώ για μία αρπαγή, για μία ε, πνευματική κλοπή η οποία γίνεται των χώρων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κυρία Άστον τι σκοπεύετε να κάνετε ε, όσον αφορά τις, τα σήματα τα οποία κατοχυρώνουν αυτές τις επιχειρήσεις αυτά, για τέτοιου είδους φυτά τα οποία πάζουν. Κύριε, επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Άστον που είστε εδώ παρούσα στην Επιτροπή μα. Είναι ε, μπορούμε να επανέλθουμε σε κάτι άλλο λεπτομερία και να μιλήσουμε για αυτή την τραγική κατάσταση την οποία επιτομίζουμε στην IT. Η κυρία Γιώργεβα, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ επαγγελματίε σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό το οποίο συνέβαινε με αυτή, μετά από αυτή την τελευταία, το τελευταίο weekend όπου ένας λέλαπας έπληξε τη χώρα αυτή, την Αϊτή και επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετάδοση της χολέρας σε αυτή την χώρα και νομίζω πως πραγματικά αυτό είναι ένα νέο πλήγμα και κατά πόσο υπάρχει μια επίγουσα απάντηση σε σχέση με αυτό το πλήγμα ιδιαίτερα υπό το φως των συμβάντων του τελευταίου weekend. Η Λέτη Έστον έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα που είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι νέο για μένα. Έχετε θέσει το θέμα τα δύσκολα θέματα στη Δική Σαχάρα, του Σαχέλ όπου έχουμε συζητήσει ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε μεγάλη ανησυχία για αυτή την περιοχή, για όλη αυτή την περιοχή της Αφρικής καθώς επίσης και τις προκλήσεις που έχουμε σε αυτές. Έχετε αυτή τη στιγμή στη Δυτική Σαχάρα τον ΟΙΕ ο οποίος δρά επίσης και έτσι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό μεταξύ των χωρών της ΕΕ και για τη λύση την οποία μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη χώρα. Το Αφγανιστάν, το Πακιστάν. Υπάρχουν επίσης προκλήσεις, διαφορετικές προκλήσεις, αλλά σημαντικές και εκεί προκλήσεις. Είναι πολύ καλό λοιπόν να βλέπει κανείς ότι την εργασία την οποία επιτελούμε ιδιαίτερα με τις γυναίκες του Αφγανιστάν, στο Αφγανιστάν είναι εκπληκτικές ότι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, σε οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξη είναι αυτή. Και στο Πακιστάν, όπως ξέρετε, εγώ είμαι προεδρεύωση της Επιτροπής εκεί η οποία ασχολείται με την κυβέρνηση η οποία βρίσκεται ενώπιον δύσκολων καταστάσεων λόγω των πλημμυρών που έχουν συμβεί. Επίσης το Αιγεμέν που αναφερθήκα. Ξέρετε αυτή είναι μια χώρα το Αιγεμέν που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα οι συζητήσει μεταξύ εντό τη χώρα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μέλη γενέστε σε αυτή τη χώρα και εργαζόμαστε σε αυτόν τον τομέα επίση. Επίση, μπορείτε να προσθέσετε το Σουδάν, τη Σομαλία και άλλε χώρε, οι οποίε όταν κοιτάτε γύρω από τον κόσμο τι γίνεται, αυτά είναι μεγάλε προκλήσει για μα, οι οποίε θα πρέπει να τι λύσουμε. Ποιε είναι οι ποιοι είναι οι πόροι του οποίου έχουμε και πώς πραγματικά θα είμαστε αποδοτικοί. Ε, οι ειδικοί εκπρόσωποι που άκουσα να λέει αναφέρεται εδώ είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω είναι άνθρωποι οποίοι είναι πάρα πολύ ε, ικανοί σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και έχουν διοριστεί και αυτό το λόγο. Σουδα, το Σουδάν, παράδειγμα. Ωστόσο, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τους βάλουμε μέσα ανθρωπιστική βοήθεια, πώς μπορούν πραγματικά να είναι καλύτεροι εκπρόσωποι για αυτό το θέμα και να διασφαλίσουμε ότι την σωστή πολιτική και με τους πόρους που διαθέτουν. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να ξανασκεπτόμαστε όλα τα θέματα αυτά εξ υπαρχής και προσπαθούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχετε δίκιο όμως ότι θα πρέπει να πάμε και αλλού και να ενισχύσουμε επιτόπου τις αντιπροσωπήσεις οι οποίες έχουμε στείλει εκεί. Το κάνουμε αυτό στο Αφγανιστάν, μπορούμε να το κάνουμε και αλλού. Και είναι σημαντικό θέμα αυτό. Κύριε Γκράτσα, αυτή τη στιγμή, όταν έγραψα, όταν μου γράψετε μάλλον για το ενδιαφέρον το οποίο έχετε, και τότε μόλις κατάλαβα τι είναι αυτό το θέμα το οποίο δεν θέλω πραγματικά να υποσπίουμε για αυτό το θέμα, διότι δεν υπήρχε όντω. Και ευελπιστούσα ότι το σκεφτήκατε αυτό το θέμα διότι γοητεύομαι, με γοητεύει αυτό το θέμα. Πάει στην ουσία του θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι πολύ ψηλά στην δική μου ατζέντα. Από άλλη σκοπιά όμως είναι ένα πολύ σημαντικό ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέματα Χρειαζόμαστε εμπεριγνώμενες σε αυτό το θέμα, αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ότι μας γράψετε για αυτό το θέμα, να μας το υπενθυμίσετε και τη δική σας, με τη δική σας συμβολή μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά σαφώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται και θα φτάσουμε ενώπιν δυσκόλων καταστάσεων. Κύριε Κάτσου τώρα, Κάτσου, για την IT. Ε, υπάρχουν δύο αρχηγοί αντιπροσωπεών που πήγαν εκεί, που βρίσκονται εκεί μάλλον. Όχι μόνο πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί ζουν εκεί, είμαστε βέβαιοι τώρα ότι ζουν αυτοί, αλλά ξέρετε ζουν με σκληρές συνθήκες, με κάτω από τις Υπάρχει προσωπικό τη ΕΕ και προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εξασφαλισμένη τροφοδότησης ένας σκοτώθηκε κιόλας. Επίσης προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία που δίδουμε να βοηθώντας αυτή την έκτακτη περίπτωση και εν τελική, αναλύση θα αποφύγουμε το χειρότερο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί φρικτά αποτελέσματα εκεί. Η κρυσταλλίνα έχει ξεκινήσει προσπάθεια και εμείς προσπαθούμε περαιτέρω να υπάρχουν περαιτέρω πόροι, περαιτέρω τέντες για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν ιδιαίτερα τα παιδιά, τα μωρά και αυτό θα, ε, θα γίνει το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαρούντα παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, λέει Άστον. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, είχαμε εκφράσει τι ανησυχίε μα για του κινδύνου, ε, τα θέματα τη ανάπτυξη να περιθωριοποιηθούν ή να τα καταπιεί η προβληματική τη ασφάλισης εξωτερική δράση. Ευχαριστώ που μα κατησυχάζετε. Άλλη ανησυχία μα είναι η σχέση τη Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης με τους ε, εθνικούς ε, υπουργούς ανάπτυξης. Οι υπουργοί αυτοί θα πρέπει να μειώσουν την παρουσία τους επιτόπου προκειμένου να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ποια είναι η άποψή σας. Υπάρχουν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις και να ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι οι 27 διαφορετικές εθνικές ταυτότητες θα είναι παρόλα αυτά παρούσες. Thank you very much, Madam President. Um, uh, Lady Ashton. Καλώς ήρθατε, Lady Ashton. Εμείς που ήμασταν στη Νέα Υόρκη για τους στόχους της κυριωτίας μπορούμε, μπορούμε να πούμε ότι οι ομιλία σας ήταν πολύ καλοί. Αν ήσασταν νευρικοί πριν έρθετε, <laughs> να σας ε, ε, πω, να σας διαβεβαιώσω ότι η δική μας ε, προσέγγιση είναι πολύ θετική απέναντι σας, παρόλο που μπορεί να είμαστε επικριτικοί που και που. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για την περιοχή του, ε, της του Σουέζ. Μιλήσαμε για το Σουδάν, για το Τζιμπουτί, για την Ιεμένη, του βομβαρδισμού στην Ιεμένη κλπ. Ας μην τα αναφέρω όλα αυτά τα κράτη. Πάντω η κατάσταση χειροτερεύει εκεί κοντά στο Σουέζ. Το δείχνει πόσο δύσκολη είναι η αποτελεσματική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς περιοχές που έχουν και κλπ. Η ερώτηση είναι, ίσω δεν έχετε βέβαια τι δυνατότητε, αλλά εσείς έχετε κάποια σύνδεση με, το, με τις στρατιωτικές δυνάμεις, με τις ένοπλες δυνάμεις ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, γιατί αυτό που κάνουν οι ένοπλες ε, δυνάμεις ενδεχομένως μερικές φορές να αντιβαίνει έμεσα ή άμεσα με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ως αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε λοιπόν με το στρατό των κρατών μελών. Ευχαριστώ Λεδιάστον. Νόιζερ. Oh, äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε Lady Άστον. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις αφήσεις δηλώσεις που κάνατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δεσμεύσεις σας σε ό,τι αφορά τις αρχές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πρόβλημα στην Βυτική Σαχάρα, γιατί υπάρχουν διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέρος αυτό. Είμαι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για την Βυτική Σαχάρα, που περιλαμβάνει περίπου 60 ε, βουλευτές του Κοινοβουλίου και να είσαστε βέβαιοι ότι είμαστε πάντα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δυτική Σαχάρα. Υπάρχει μια άσχημη εξέλιξη. Σήμερα υπήρξε επιτρομή ε, μαροκινών δυνάμεων στην, στα κέντρα ε, όπου στεγάζονται 12.000 άτομα και ένας ε, νεαρός 14χρονος σκοτώθηκε. Σας ρωτώ λοιπόν ποια δέσμευση θα αναλάβουμε. Ξέρουμε ότι η ΟΗΕ έχουν, έχει αποστείλει πρεσβευτή επιτόπου αλλά θα έπρεπε να ε, δείξει μεγαλύτερη πυγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Κύριε Σπένσον, χαίρομαι που καταλαβαίνετε πως ε, η αναπτυξιακή πτυχή ε, δεν θα καταβαραθρωθεί και αυτό θα φανεί σύντομα, σιγά σιγά. Ρωτήσατε όμως για την σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επιτόπου με τη δράση των 27 κρατών μελών. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι ε, να συντονίζει τα κρατη επιτόπου. Όχι να ελεπικαλύπτεται με τα κράτη-μέλη, αλλά να παρέχει δύο πράγματα. Πρώτον, να εξασφαλίζει μια συνέπεια ε, και λογική συνέχεια του μηνύματος που βγαίνει προς τα έξω Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι και δεν είναι 27 παρόντες βέβαια, είναι 3, 4, 5 χώρες. Ε, και δεύτερον, όταν κάποιος ε, πάει σε μια πρεσβεία κάπου στον κόσμο, ε, πάντοτε ξέρει σε ποια χώρα βρίσκεται. Όταν όμως πάει στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρει, πρέπει να ξέρει. Και θα πρέπει η δική μας παρουσία εκεί να είναι παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δίνει μια ταυτότητα ευρωπαϊκή στην παρουσία μας. Συνεπώς, συνεργαζόμαστε, συντονίζουμε, δίνουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα στην παρουσία μας, αλλά δεν αλληλεπικαλυπτόμεθα με τα κράτη-μέλη, ούτε και τους αφαιρούμε δυνατότητα δράσης. Το αντίθετο. Το κ. Νιούτοντον Το θέμα της διόργας του Σουέζ ασφαλώς και μας απασχολεί. Αν δείτε τις ε, γειτονικέ χώρες θα διαπιστώσετε πράγματι πολλά προβλήματα. Το ερώτημα είναι πώς αυτό που κάνουμε σε ένα τομέα, σε ένα πεδίο δεν ε, θα επηρεάζει αυτό που κάνουμε σε άλλα. Θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία Αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περιοχή δεν συμπληρώνουν ή δεν συμπληρώνονται από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες περιοχές. Το αντίθετο μάλιστα μερικές φορές. Και η Λισαβόνα θα βοηθήσει αυτό. Θα μας βοηθήσει όλα τα κομμάτια του παζλ να είναι το ένα δίπλα στ' άλλο. Να ταιριάξουν έτσι ώστε η ανταπόκρισή μας να ε, είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Η συνεργασία με το στρατό, για παράδειγμα στην ΑΕΤ, ήταν εξαιρετικά σημαντική, ζωτική σημασία. Γιατί ο στρατός δεν ήταν εκεί ο στρατός, ο στρατός ήταν εκεί επειδή έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις κρίση πολύ γρήγορα. Μερικέ ε, φορέ οι στρατιωτικέ μα δραστηριότητε όμω αφορούν την ασφάλεια μια συγκεκριμένη χώρα. Και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην εξασφάλιση ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως θα πρέπει η στρατιωτική παρουσία να είναι συμπληρωματική. Συνεργάζομαι με τους, ε, ε, τα σημεία επαφής των, τους, των όπλων δυνάμεων των διαφόρων κρατών μελών και επίσης έχουμε βέβαια και Συμβούλιο Υπουργών, όπως έχουμε Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης από κοινού. Τώρα, για τη Δυτική Σαχάρα. Τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες η Δυτική Σαχάρα ε, ήταν στο προσκήνιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη. Πλην όμως <laughs> αυτό δεν μου είχε, αυτό δεν το είχε προβλέψει κανένα σε μένα τουλάχιστον. Ε, δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μία, ένα, μία κοινή ε, στάση. Βέβαια τα Ηνωμένα Έθνη ηγούνται της προσπάθειας. Μπορώ να το συζητήσω με τα Ηνωμένα Έθνη. Το πρόβλημα βέβαια, σας επαναλαμβάνω, ότι δεν έχουμε κοινή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξεπεράσω αυτό το ζήτημα. Θα το δω με τον Οργανισμό Εθνών. Είναι πάρα πολύ δυσχερή η κατάσταση εκεί για τους κατοίκους και πρέπει να το ξαναδούμε. Thank you very much. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε πολύ ορθώς ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι που πάνε τα χρήματα και ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Συμφωνώ. Αναρωτιέμαι όμως γιατί κονδύλια διατίθενται για παράδειγμα για τη Frontex ή γιατί διατίθενται κονδύλια ε, στη Συμφωνία Πλαίσια για τη Λιβύη. Δεν είμαι βέβαιη τι κάνουν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά, αλλά σίγουρα δεν βοηθούν στην εξάλληψη της φτώχειας. Να ρωτήσω όμως σε ό,τι αφορά τα πολιτικά θέματα, τα θέματα πολιτικής για τα ζητήματα αναπτυξιακής βοήθειας. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα προωθήσει και θα διασφαλίσει το PCD και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στο εμπόριο, και πώς θα διασφαλίσετε ότι υπάρχει συμφωνία αναπτυξιακή εντός της υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την τεχνοσία. Και τέλος, πώς θα διασφαλίσετε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εξωτερικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαι βέβαιη ότι είσαστε απόλυτα δεσμευμένοι για τα θέματα αυτά. Αλλά ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν ότι όλοι θα συμφωνήσουν με τη δέσμευσή σας και θα παραμείνει αυτή η δέσμευση στη θεωρία, αλλά αφαιρεθεί σε πράξη. Συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ευχαριστώ, η ε, κυρία Χούλη. Ευχαριστώ. Για να επανέλθω στο θέμα, σε αυτό που είπατε για τον κύριο Μπένσον, ως απάντηση στον κύριο Μπένσον, όταν ήμουνα η επικεφαλής της ομάδας στη Μοζαμβίκη, Κάτι που με έκανε εντύπωση ήταν ότι είχαμε 15 επικεφαλής αντιπροσωπιών, 15 κράτη-μέλη εκπροσωπούντας τη Μοζαμβίκη. Και αναρωτιόμουν σε συνθήκες, συνθήκες πίεσης, όπου οι προπολογισμοί των κρατών μελών είναι υποπίεση. Θεωρείτε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν ανοίγει μια δυνατότητα να εξοικονομήσουν κάποια τέτοια έξοδα τα κρατημέλη, μειώνοντα την εκπροσώπησή του στο εξωτερικό και θα υποστηρίξετε, θα ενθαρρύνετε τα κρατημέλη και το δικό μας κράτος να προβούν σε τέτοιες οικονομίες. Μας δίνει λίγο χρόνος, λίγο ακόμη και θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη εταιρεσκερός γύρος, εάν θέλετε, για αυτές τις ερωτήσεις οι οποίε ετέθησαν. Χωρί μικρόφωνο δυστυχώ ο μιλητής, χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούμε τίποτα. Ναι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή μονάδα η οποία θα είναι επίσημη για να παρακολουθεί με τη συμμετοχή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί μαζί με την Κομισιόν τη εξωτερική προσπάθεια την οποία κάνουμε για να γίνει ένας απολογισμός όσον αφορά αυτή την εξωτερική βοήθεια και να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσει στους στόχους που έχουν τοθεί και δεύτερον να συζητάει στα πλαίσια της δικής μας Επιτροπής με το πέρας της πρώτης ε, χρονιάς τα αποτελέσματα. Το επαναλαμβάνω αυτό το αίτημά μας. Δεν βεβαίως αυτή τη στιγμή να κάνω έναν, μια δίκη ε, κατηγορώντας ότι δεν θέλετε να το κάνετε κάτι τέτοιο. Πλην όμως πρέπει να σας το υποβάλω για δεύτερη φορά αυτό το αίτημα. Η ας τον έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα το οποίο θέσατε είναι δική μας εξωτερική δραστηριότητα και είναι δική μου. Νομίζω πως πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα τα μέλη του Κοινοβουλίου εδώ, του σώματος αυτού, να νιώθουν, να αισθάνονται μέλη αυτής, αυτής της προσπάθειας, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη δέσμευση την οποία έχει αναλάβει αυτή, αυτή η Επιτροπή και κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα έχουμε αυτά αποτελέσματα και η προσπάθειά μας θα είναι πάρα πολύ σημαντική για να επιδειχθεί αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Το εμπόριο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλές χώρες και νομίζω πραγματικά η δυνατότητα να εμπορευόμαστε με αυτές τις χώρες ήταν, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να υπάρχουν δημιουργώντας αυτό το διάδρομο νοραβό του νο, ε, <laughs> βορρά νότου κλπ. Πράγμα το οποίο άπτεται βεβαίω τον υπόδο και σε αυτόν τον τομέα έγιναν πολύ σοβαρέ εργασίες για να αναπτύχθει η οικονομία τους και κάτι άλλο το οποίο είναι απολύτω σημαντικό για μένα να το πω για την εξαγωγή των πρώτων υλών. Εγώ το για τις χώρες οι οποίες εξάγουν μάγκο, για παράδειγμα το προϊόν το φρούτο, ξέρετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται οικονομικά όπου φτιάχνουν το chutney, μια σάλτσα αγγλική από το μάγκο και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να αναπτυχθούν, να το εξάγουν καλύτερα και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ αυτών των πραγμάτων και της ανάπτυξης η οποία προκύπτει εκεί. Έτσι λοιπόν εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα στην ανάπτυξη. Επίσης οι μηχανισμοί είναι, κάτι, η ουσία του πράγματος. Μπορούμε να δώσουμε γραμμές, οδηγίες, κατευθύνσεις, κατε... αλλά το πιο σημαντικό είναι και το οποίο λέγεται αυτή τη συνθήκη είναι πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το πράγμα και αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε προσπάθειάς μας. Βεβαίως έχουμε εμπο... Ε, πρεσβευτές, έχουμε αρχικούς των αποστολών, όχι μόνο αυτών, αλλά θα πρέπει να γίνεται μέσα από ομάδες management διαχείριστης και είναι κάτι δικό μου που κάνουμε, η δική μου υπηρεσία και αυτό είναι το, η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στους μηχανισμούς που, οι οποίοι υπάρχουν. Κύριε κυρία μίλησε για τη Μοζαμβίκη. Μειώνουμε λέει αυτή τη στιγμή, όχι όχι, τζόκι, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν μειώνουμε τις αντιπροσωπείτες. Ότι υπάρχουν αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται και είναι κυρίαρχε αποφάσει που λαμβάνονται από ορισμένε χώρε. Αλλά αυτό δεν αποτελεί ένα, μια δικαιολογία για να γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό που πήγαμε εμεί να κάνουμε σαν Ευρώπη εκεί θα πρέπει να λειτουργεί στον κόσμο και βεβαίω δεν είναι αυτό μια δικαιολογία για τα κράτη-μέλη να αποφεύγουν να κάνουν τη βοήθεια που πρέπει να κάνουν. Είμαστε αποφα... Είμαι αποφασισμένη και εγώ προσωπικά να μην υπάρχει υποκατάστατο, αλλά να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας εκεί όπως πρέπει. Κύριε Κέρντς, δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσον ε, αυτό το θέμα των, της διαμάχης είναι αλήθεια. Νομίζω πως πραγματικά θα πρέπει αυτή η Επιτροπή να δει τα θέματα αυτά, να τα συζητήσει εδώ και συγγνώμη και θα καταλάβετε το γιατί, διότι δεν πρέπει να επιμένουμε στις διαμάχες που δημιουργούνται. Η Κρυσταλίνα και εγώ συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε κάτι καινούριο και προς το παρόν δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε τη λύση σε αυτό το θέμα και να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε αυτό, θα κατορθώσουμε να μην υπάρχουν διαμάχες όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Κύριε Κάιζερ, έχετε ξανά το λόγο. Έχω τύψεις, κύριε Άστον, για να επανέλθω στο ερώτημά μου, διότι δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, σε μηχανία και καταλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και το είπατε εσείς και στις απαντήσεις οποίες δώσατε, όταν βλέπετε τη σημασία που έχουν αυτές οι, αντι, αντιπροσωπείες για τον έλεγχο των εξετάσεων και δεν ξέρετε όλα τους μηχανισμούς και όλα τα όλο το, μηχανισμό που ζητούργει. αλλά ωστόσο υπάρχουν πολλές αποστολές στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν λοιπά, είναι διαφορετικού τύπου και σε ένα ορισμένο, σε ένα ορισμένο βαθμό η ΕΕ και οι ΟΗΕ συνεργάζονται πολύ στενά και βεβαίω ο ΟΗΕ υποστήριζε την έψινεψη. Στο, Σουδάν, στο Σουδάν όμως άλλαξε η πολιτική και άλλαξε η πολιτική σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λέει πανέ ότι δεν θα υπάρχει δεν πρέπει να υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των αντιπροσωπιών οι οποίες είναι για τη διασφάλιση της ειρήνης και ημών. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Δεν θα πρέπει να πούμε ότι να κάνουν όλη αυτή την υποστήριξη να είναι το δίκτυο προστασίας αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε να υπάρχουν άλλες διατάξεις και άλλες αποφάσεις που να ληφθούν θα μιλήσετε με τον ΟΗΕ θα μιλήσετε για το Δυτική Σαχάρα ναι και εάν πραγματικά ο καθένας προωθεί τα δικά του πιόνια δεν αρκεί πρέπει να μιλήσουμε με τον ΟΗΕ να υπάρχει μια συνεργασία για να διευκρινιστεί και να διασφαλιστούν αυτές οι αποστολές εκεί και αλλού. Δεν θέλω όμως να σας πιέσω, καταλαβαίνω ωστόσο είναι παιδεία τα οποία είναι λίγο θα λέγαμε ναρκοθετημένα εν μέρη προς σε σχέση. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε, για τον τρόπο που προεδρεύσατε εδώ πέρα στην ε, συνεδρίαση, γιατί πολλά μέλη θέλουν να θέσουν ερωτήσεις, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και χαλαρή η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Άστον που μας αφιέρωσε το χρόνο αυτό και λέγοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, γιατί ασχολούμαστε και με τα καινούργια προβλήματα που ανακύπτουν και η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη φυσικά από τη θεραπεία. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζω και τα οποία δεν έχουμε ακόμα θίξει είναι οι 300 ε, λίμνες που έχουν σχηματιστεί γύρω από τα Χιμαλάια και οι οποίες είναι έτοιμες να ε, ξεχυλήσουν. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία του ICI. Υπάρχει λοιπόν τήξη των πάγων ε, στα Χιμαλάγια η οποία επιταχύνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμέναμε λόγω του άνθρακα. Δεν έχει να κάνει με την ε, παγκόσμια θέρμανση, με τη θέρμανση του κλίματος. Δεν συζητήθηκε στην Κοπεχάγη, μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει θίξει το θέμα αυτό. Επέστρεψε και μόλι ο συνάδελφο από το Κατμαντού. Πέταξε σε 1800 μέτρα ύψος με ελικόπτερο και μας αναφέρει το τι γίνεται εκεί πέρα. Πρόκειται για μια επικείμενη καταστροφή. Οι ποταμοί υπερχιλίζουν και οι ποταμοί αυτοί, ξέρετε, ε, θρέφουν 1,2 δισεκατομμύρια κόσμο και όλα αυτά πλέον διακινδυνεύονται. Όχι λόγω της ε, θέρμανσης του κλίματος, αλλά λόγω του μαύρου άνθρακα. Έχετε λοιπόν κάτι επιπλέον για να ανησυχείτε, πέρα από τη Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Λέει Άστον, έχετε το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να κάνετε κάποιες και τελικές παρατηρήσεις ενδεχομένως αν θέλετε. Δεν έχω να σας δώσω απάντηση για το δίχτυ ασφαλείας. Ακόμα. Ε, κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε ως τώρα. Τις τελευταίες τρεις ε, μέρες δεν μου έχουν πει τι έχει γίνει. Πλην όμως ξέρω ότι γίνονται πράγματα. Θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα δίκτυ προστασίας. Σας είπα και προηγουμένως, η ασφάλεια είναι ζωτική σημασία. Νούμερο ένα. Θα το δω. Σε ό,τι αφορά τις λίμνες στα Ιμαλάια. σε κάτι συνεδρίες κάτι μαθαίνω, το λέω. για παράδειγμα, για την βιοπειρατεία. Έμαθα λίγο πριν έρθω. Τώρα μαθαίνω και για αυτό το πρόβλημα. και δεν την πιστεύω τα αυτιά μου. Δεν έχω ιδέα για το ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι λύσεις. Λέτε ότι οφείλεται στην εθάλη και όχι στο, στο, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Θα το δω. Λοιπόν, ε, ως τελικές παρατηρήσεις να ευχαριστήσω την κυρία Ζολή για την ευκαιρία που μου έδωσε. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ μας, ε, με βοήθησε σε πολλά σημεία. Πρώτον, βλέπω τη σημασία που την Επιτροπή στην ε, αποτελεσματικότητα των δρασιών μας. Επιθυμεί η Επιτροπή τα θέματα ανάπτυξης να βρίσκονται στην καρδιά της δράσης μας. Αλλά συμπληρωματικά. Συνεπώς δεν θα πρέπει απλώς να συνδυάσουμε τα διαφορετικά γρανάζια της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να αποφύγουμε επιτόπου κατά τη στιγμή της δράσης να ερχόμαστε σε συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό το πρόβλημα που χρειάζεται να σκεπτόμαστε κάθε φορά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με πιο ευφύ τρόπο. Με καινοτόμη, καινοτόμη χρηματοδότηση, με συνεργασία, με αναγνώριση ότι οι προκλήσεις γίνονται όλο και πιο ε, μεγάλες, πιο σημαντικές, με την πρόληψη, με την πρόβλεψη που θα δημιουργηθούν προβλήματα κλπ. Επαναβεβαιώσαμε σήμερα ότι η συνθήκη της Λισαβόνα μας δίνει μια πραγματική ευκαιρία να δράσουμε καλύτερα, να πετύχουμε περισσότερα, να μείνουμε πιστοί στο όραμά μας και καταλαβαίνω την ανησυχία σας ε, εν το μέσο οικονομικής κρίσης τα θέματα ανάπτυξης να μην επισκιαστούν θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να εξασφαλίσουμε διαφάνεια, να αποδεικνύουμε τι κάνουμε και για ποιο λόγο το κάνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα η επιτροπή αυτή είναι το σημείο στο οποίο ο Άντρης, η Κρυσταλίνα και εγώ θα μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα, να μάθουμε. Έμαθα πολλά πράγματα σήμερα ήδη. Και βλέπω ότι αυτό είναι, επιτελείται πολύ σωστά το ρόλο σας. Είμαι περήφανη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρου τη Επιτροπή, ευελπιστώντα ότι πραγματικά αυτή η παρουσίαση εδώ θα είναι τήσια. Άρα θα σα δούμε την επόμενη χρονιά. Καλή τύχη για την εκτέλεση των εργασιών, καθώ επίση και την επιτέλεση του έργου σα, το, του έργου το, το οποίο έχετε αναλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat>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 Nous allons reprendre notre réunion et le point 7. Περνάμε στο σημείο Μάλλον, συγγνώμη, επιστρέφουμε στο σημείο 7 της Μέσιας Διάταξης, διότι δεν το είχαμε ολοκληρώσει. Δίνω το λόγο ξανά στη Μισελ Στρίφλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρουσίασα την έκθεσή μου. Θα ακούσω τώρα από εσά προτάσεις ή ερωτήσεις. Δεν ξέρω πότε είναι η ερωτήσει. δεν ξερω ποτε ειναι η προθεσμια για την υποβολή τροπολογιών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς καταρχήν. Ε, μιλούμε για την... Μιλούμε για την συγγνώμη, δεν, άκουσα τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί μιλάμε, ε, γιατί έχει πολύ θόρυβο η αίθουσα. Ε, λέει η κυρία Στρίφλερ, είχα παρουσιάσει την έκθεσή μου, την είχαμε διακόψει, οπότε τώρα περιμένω από εσά σχόλια. Έχω μια πρόταση, λέει ο κ. Γκέρνς. Με την Επίτροπο, την κυρία Γεωργίεβα, συζητήσαμε το θέμα της μελλοντική ε, χρηματοδότησης των δράσεων στον τομέα της. Ε, το Ταμείο σχεδόν άδειο. Οπότε δεν πρέπει να γίνει καμία καταστροφή, καμία θεομηνία από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουμε πώς να χρηματοδοτήσουμε την ανθρωπιστική δράση Οπουδήποτε. Πια. Αναζητούμε λοιπόν δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας, ε, από κοινού συνεργασίας, από κοινού χρηματοδότηση κρατών μελών και κομισιών. Και αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν δράσεις τις οποίες θα διαχειρίζεται και θα φέρει πέραση κυρία Γεωργίεβα Δηλαδή, δράσεις οποίες, τις οποίες θα έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη ε, μετά βέβαια από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα ο κάθε, κάθε χώρα έδινε τον οβολό της ε, με την ευκαιρία μια της α ή της β καταστροφής αλλά χωρίς συντονισμό και χωρίς ε, να ε, υπάρχει μια γενικότερη, ένας γενικότερος συντονισμός. Συνήθως, σε περίπτωση ανεπάρκειας πιστώσεων, ίσως θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη χρημάτων, αλλά και την έλλειψη συντονισμού. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Στρίφλερ. Uh, Ένα-δυο σχόλια από την πλευρά της Κομισιόν. Καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση ιδιαίτερα επειδή θέλει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μιλάει επίσης για τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ε, σημασία του να φτάσουμε στους ανθρώπους που πλήττονται κάθε φορά. Επίση η εκθεσή σας μιλάει για τις διεθνεί κατευθυντήρε γραμμέ που για μα είναι πολύ σημαντικέ επίση. Ω απάντηση στον κύριο Γκέρεντς ε, και εμείς ε, θα συμφωνούσαμε να συμπληρωθούν τα ποσά που διαθέτουμε εμείς με ε, από τα κράτη-μέλη. Παλαιότερα, κράτη-μέλη μας είχαν... Ε, μάλλον είχαν αιτηθεί να δαπανούμε εμείς ποσά εξ ονόματός τους εκ μέρους τους. Όμως, ε, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτό δεν είναι δυνατό. Ε, το 2011 το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν προβλέπει αναθεώρηση αυτού του κανονισμού, οπότε ενδεχομένω θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και αυτό το θέμα στην αναθεώρηση. Η έκθεση δίνει σημασία και στο θέμα της κοινή ε, ευρωπαϊκής αντίληψης και της ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί και εμείς εργαζόμαστε και με τα κρατημέλη και με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της ορατότητας, της κοινή αντίληψης σε εθνικό επίπεδο. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στις διμερείς μας επαφές με το Συμβούλιο και, με... και το... η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου το υπογράμμισε. Ε, προσπαθούμε σε αυτές τις επαφές να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ορατότητα της κοινή αντίληψης στα κράτη-μέλη. Και ένα σχόλιο. Πολύ σωστή είναι η υποστήριξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και η πρόθεσή του. Δεν είμαι σίγουρη όμως για το αν θα έπρεπε να, αυτό να γίνει με κονδύλια από την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τη Διεθνή Επιτροπή Ερθρού Σταυρού για την πρόθεση του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά γίνεται και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται με χρηματοδότηση από άλλα κεφάλαια του προπολογισμού της Κομισιόν, διότι δεν έχουμε ε, περίσευμα ε, πόρων ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης θα θυμάστε ότι ετοιμάζουμε μια ανακοίνωση για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση ε, του, της κοινή αντίληψης. Εκεί θα συμπεριλάβουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη τους τρεις-τέσσερις τελευταίους μήνες, γιατί είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Συνεπώς εκεί στην ανακοίνωση θα αναφέρουμε και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης μέχρι τώρα επί, την, επί τη βάση των πληροφοριών που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Θα τα λάβω υπόψη αυτά που είπατε, λέει η κυρία Στρίφλερ. Να σας πω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου και προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 17 Νοεμβρίου. Περνάμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης. Φορολογία και ανάπτυξη. Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα. Ήδη σας είχα παρουσιάσει προφορικά αυτήν την έκθεση στην προηγούμενη μας συνάντηση. Σήμερα λαμβάνει η χώρα η δεύτερη ανταλλαγή προφοριών. Η έκθεση αυτή δεν έχει μεταφραστεί, βρίσκεται μόνο στα αγγλικά. Συνεπώς θα συνεχίσω τις συζητήσεις για αυτό το θέμα στα αγγλικά. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ε, προτάσεις για να υποστηριχθούν οι απόψεις κομισιών για το θέμα αυτό και να την ενθαρρύνουν να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αναγνώριση ε, της επιτυχίας των, ε, της σχέσης ανάμεσα στην επιτυχία των στόχων της χιλιετίας και των, της φορολογικής διακυβέρνησης η συμμετοχή, συμπερίληψη αυτών των θεμάτων στα έγγραφα τα σχετικά με τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου και τα διάφορα κράτη. Η σημασία των συμφωνιών ανταλλαγής προλογικών ε, δεδομένων στο πλαίσιο συμφωνιών με τα, διάφορα ανσόμενα κράτη κλπ. Δεύτερο σημείο, υπάρχουν προτάσεις ε, για την υπογράμμιση του αρνητικού ρόλου των φορολογικών παραδείσων που ε, οξύνουν τα φορολογικά προβλήματα, τα δημοσιονομικά προβλήματα των ψώμων χωρών. Γιατί μειώνουν το φορολογικό ε, ανταγωνισμό και δίνουν ιδιαίτερους υπερβολικά ευνοϊκούς όρους για να προσελκύσουν κεφάλαια. Η φορολογική παράδειση αυξάνοντας ε, τον ανταγωνισμό για την ε, προσέλκυση κεφαλαίων υποσκάπτουν το, την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών που ήδη έχουν μικρή φορολογική βάση. Οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες δίνουν ε, φορολογικές ελαφρύνσεις σε μεγάλες ε, εθνικές και ξένες εταιρείες προκειμένου να προσελκύσουν, ε, προσελκύσουν επενδύσεις. Ο φορολογικός ανταγωνισμός μετακινεί το φορολογικό βάρος σε χαμηλοεισοδηματίες και εργαζόμενους. Και αυτό βέβαια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες σε αμψόμενες χώρες. Τέλος, έχουν γίνει προτάσεις των πρασίνων για να αντιμετωπίσουν ορισμένε αδυναμίε τη ανάλυση Κομισιών που έχουν σχέση με τι εξή ιδέε. Η Κομισιόν δεν αναφέρεται στον αρνητικό αντίκτυπο της ε, απελευθέρωσης του εμπορίου και της μείωσης των δασμολογικών εσόδων. Στην έκθεσή μου θα υπογραμμίσω την μείωση των ε, εμπορικών φόρων που προκύπτει από περιφερειακές συμφωνίες και από συμφωνίες του ΠΟΗ και θα αναδείξω το γεγονός ότι αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις φτωχότερες χώρες που έχουν χάσει το 30% των φορολογικών του εσόδων εξαιτία αυτών. Η Κομισιόν δεν κάνει προτάσεις για την διεύνηση φορολογικής ε, βάσης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα ε, πιο δίκαιο ε, φορολογικό σύστημα. Οι πράσινοι προτείνουν ε, να πούμε ότι η μείωση των φορολογικών ε, εσόδων έχει οδηγήσει σε αύξηση των φόρων κατανάλωσης, όπως ο ΦΠΑ ας πούμε. Όμως παρόλο τη διεύρυνση που προκύπτει, της φορολογικής βάσης προκύπτει από τον ΦΠΑ δεν είναι το κατάλληλο μέσο διότι πλήττει πιο πολύ τους πιο φτωχούς. Συνεπώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθεί στην ανάπτυξη των συστημάτων άμεση φορολόγηση στι αναπτυσσόμενε χώρε. Οι αναπτυσσόμενε ε, χώρε ε, χρειάζονται, χρειάζεται να μπορούν να εφαρμόσουν ε, μέτρα ελέγχου των κεφαλαίων για να αποφύγουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν σταθερότητα. Η Κομισιόν θα πρέπει να υποστηρίξει τι αναπτυσσόμενε χώρε στην προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα, στα διεθνή φορολογικά πρότυπα. Όμως, η Κομισιόν δεν επικρίνει καθόλου τι ε, αδυναμίες του ΟΣΑ αυτή τη στιγμή. Ο κώδικας του ΟΣΑ επιτρέπει σε διάφορες χώρες να ξεφύγουν υποσχόμενες ότι στο μέλλον θα συμμορφωθούν με τους κανόνες. Ε, ο τρόπος να διαγραφούν από το μαύρο κατάλογο είναι να συνάψουν 12 συμφωνίες με άλλες χώρες χωρίς όμως να έχει αξιολογηθεί αντικειμενικά σε κάθε περίπτωση η συμμόρφωση με τους κανόνες καλής διακυβέρνησης. Χρειάζεται ο κώδικας του ΩΣΑ ε, προβλέπει ανταλλαγή στοιχείων κατόπιν αιτήματο, αλλά όχι αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων. Και βλέπουμε ότι η φορολογική παράδειση αρχίζουν και συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους προκειμένου να βγουν από το μαύρο κατάλογο. Ε, αυτό όμως προφανώς ε, δεν λύνει το πρόβλημα. Οπότε προτείνουμε να να πάμε πιο μακριά από τον κώδικα του ΩΣΑ, να ζητήσουμε μια διεθνή σύμβαση με στόχο να καταργηθούν τέτοιου είδους βλαβερές φορολογικές ε, πρακτικές ε, και να ε, επιβληθούν αυστηροί όροι στις εταιρείες που δρούν σε φορολογικούς παραδείσους. Η Κομισιόν ε, δεν σχολιάζει το θέμα του πόσο οι φορολογικές συμφωνίες ε, βοηθούν στην ανάπτυξη φορολογικών, καταλο... ε, φορολογικών παραδείσων. Συνέπως εμείς ως ε, πράσινοι θεωρούμε ότι οι εταιρείε θα πρέπει να φορολογούνται με βάση τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες χώρες όπου δραστηριοποιούνται και όχι εκεί που είναι εγκατεστημένη η έδρα τους. Η Κομισιόν Ε, αναφέρει την αρχή arm's length αλλά δεν προτείνει άλλες μεθόδους. Εμείς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην χρήση ε, διαφόρων κανονισμών για την, ε, τον εντοπισμό ε, λανθασμένης τιμολόγησης των συναλλαγών. Για παράδειγμα, ε, μεθόδους συγκρίσιμου κέρδους. Οπότε προτείνουμε ε, να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις έτσι ώστε η G20, ο ΣΑΤ, ο ΙΕ ε, και ο ΠΟΕ να καθορίσουν ένα πιο ευρύ κατάλογο κριτηρίων και μεθόδων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λανθασμένης τιμολόγησης των συναλλαγών. Η Κομισιόν δεν αναφέρεται επίσης στη διάβρωση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από το φορολογικό ανταγωνισμό μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οπότε προτείνουμε ή να δώσουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να επιβάλλουν ε, ελέγχους στα κεφάλαια προκειμένου να αποφύγουν ε, κερδοσκοπικές δράσεις και να εξασφαλίσουμε συμφωνίες με αυτές τις χώρες έτσι ώστε οι εθνικές ε, επιχειρήσεις και οι διεθνείς επιχειρήσεις να, θα πληρώνουν ε, επαρκείς φόρους. Αυτό είναι το περιεχόμενο ε, της έκθεσης που έχετε ήδη στο φάκελό σας. Ο λόγος σε εσάς, ο κ. Γκερέρο καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και που είσαστε και συγγήτρια ταυτόχρονα. Σε αυτή την έκθεση την οποία συζητούμε. Η έκθεσή σας ε, μας κάνει μια πολύ καλή περιγραφή και μας εξηγεί τη σημασία της ε, φορολόγησης στην επιτυχία των ε, ανησιακών μας στόχων. Η σοσιαλιστική ομάδα υποστηρίζει την ε, θέση της έκθεσης σε ό,τι αφορά την ενίσχυση υπέρ του φόρου. Δηλαδή, ε, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καταρτιστούν, να τις βοηθήσουμε να καταρτιστούν σε θέματα φορολογικής διαχείρισης, φορολογικής διοίκησης και ταυτόχρονα να εφαρμόσουν με φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάστασή τους. Διότι θεωρούμε πως ένα ευρώ που επενδύεται στην βελτίωση της φορολογικής διακυβέρνησης μπορεί να κινητοποιήσει 10 ακόμα ευρώ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ζητούμε λοιπόν από τις χώρες οι οποίες ακόμα δεν έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση αμοιβαία συνδρομής ε, για φορολογικά θέματα του ΟΣΑ να το κάνουν, να το πράξουν όχι γιατί πιστεύουμε πως είναι το, ε, το σημείο τερματισμού αλλά σίγουρα είναι ένα κρίσιμο σημείο από το οποίο πρέπει να περάσουμε όλοι. Η σοσιαλιστική ομάδα επίσης υποστηρίζει την πρόοδο στο, αυτό που ονομάζουμε country by country report, δηλαδή στις εκθέσεις που ε, ομαδοποιούν τις ε, δραστηριότητες ε, κάποιες συγκεκριμένες επιχείρησεις σε κάθε χώρα. Ζητούμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο περισσότερη δράση στο θέμα της οδηγίας για τη ε, διαφάνεια των εξορρυκτικών επιχειρήσεων. Και βέβαια η σοσιαλιστική ομάδα επίσης είναι υπέρ του αγώνα της, ε, μάχης κατά των φορολογικών παραδείσων της ε, νομοποίησης παρανόμου χρήματος και του τραπεζικού απορρίτου. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς ένα αυτό αυτόματο μηχανισμό ανταλλαγής ε, φορολογικών ε, πληροφοριών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Διεθνή Συνεργασία του ΟΗΕ ε, και θα υποβάλουμε μάλιστα και μια τροπολογία για την καλή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα, μια τροπολογία που έχει ως στόχο την υιοθέτηση μιας ε, ε, ρήτρας φορολογικής διαφάνειας ε, σε όλες τις συμφωνίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει με τρίτες χώρες. Τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι τα φορολογικά θέματα δεν σχετίζονται μόνο με κινητοποίηση πόρων, αλλά κυρίως σχετίζονται με τη σχέση ανάμεσα στην δημόσια διοίκηση και τους πολίτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα ο φόρος, είναι και ζήτημα δημοκρατίας, λειτουργίας της δημοκρατίας και βέβαια ζήτημα λογοδοσίας. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur ναι, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να σας συγχαρώ ως εισηγήτρια για την έκθεση η οποία λαμβάνει υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία, όλες τις σημαντικές πτυχές του θέματος. Είναι απόλυτα σαφές ότι κάθε κράτος μέλος και κυρίως ε, τα αναπτυσσόμενα κράτη θα πρέπει να έχουν σωστή φορολογική πολιτική αν επιδιώκει την βιώσιμη ανάπτυξη. Το, το ότι σήμερα αυτό δεν συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται εν μέρη στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, όπου και στον φορολογικό τομέα υπάρχουν ε, πάρα πολύ έντονα φαινόμενα διαφθοράς και πολλά χρήματα χάνονται αλλά οφείλεται και στις αναπτυχμένες χώρες οι οποίες αξιοποιούν όποια ευκαιρία έχουν για να μειώσουν το φορολογικό τους φόρτο. Και τεχνητά μεταφέρουν τα κέρδη προκειμένου να πληρώνουν όσο πιο μικρό φόρο γίνεται. Αυτό δεν συμβαίνει φυσικά μόνο στις ε, χώρες της αναπτυσσόμενης, συμβαίνει και στην Ευρώπη. Γιατί φυσικά στο ιστορικό της Ευρώπης, αν ε, κάποια χώρα έχει υψηλό φορολογικό καθεστώς, προσπαθούν να την αποφύγουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επί της αρχής να υπάρχει φορολόγηση όπου, γίνεται, όπου υπάρχει δραστηριότητα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει σχετικά πιο πολύ δραστηριότητα σε μία χώρη, χώρα από τη σε άλλη, αλλά μπορεί για παράδειγμα να μην υπάρχουν πολλά κέρδη στη μία από τις δύο χώρες και το καθεξής. Επί της αρχής θεωρώ ότι ο στόχος πραγματικά είναι ο εξής, να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και όσα έχει σημειώσει κάποια επιτυχία, κάποια πρόοδο. Δεν έχει φτάσει στον ε, τελικό στόχο, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα δυσκολεύουν. Η φορολογική παράδοση θα δυσκολεύονται στα επόμενα χρόνια και καλώς θα δυσκολευτούν. Και επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όντως να κοιτάξουμε την ένταση της οικονομικής δραστηριότητας και να φροντίσουμε στις μονομένες χώρες όπου λαμβάνει η χώρα η δραστηριότητα να γίνεται η φορολόγηση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ε, αναλογικά προς την ε, έκταση της δραστηριότητας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι κρύβεται και πίσω από κάθε δραστηριότητα και κάτι που θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας στα αναπτυσσόμενα κράτη χρειαζόμαστε απλά φορολογικά συστήματα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στις δικές μας εμπειρίες και να λάβουμε υπόψη τα δικά μας φορολογικά συστήματα προσπαθώντας να τα εφαρμόσουμε σε αυτές τις χώρες. Και λαμβάνοντας υπόψη και παράδειγμα τι γίνεται στη Γερμανία. Δεν είναι καλό παράδειγμα. Είναι πραγματικά πολύ εκτενής ε, ε, η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη φορολογία και κάθε κράτος μέλος αναπτυσσόμενο θα αντιμετώπιζε προβλήματα να εφαρμόσει ακόμα και το μισό από όσα ισχύουν στη Γερμανία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι το κράτος δεν θα μπορεί να βάλει χέρι στα ταμεία για να μην εξαφανίζονται σε σκοτεινά κυκλώματα τα λεφτά του φορολογούμενου. Στη Νέα Υόρκη ξέρουμε όταν συζητήθηκαν πριν από δύο ε, μήνες ε, οι στόχοι της χιλιετίας ακούσαμε ότι πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά κονδύλια χάνονται λόγω της διαφθοράς και αυτό πλήττει φυσικά και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να προσέξουμε λοιπόν. Θεωρώ ότι επί της αρχής είναι καλή η προσέγγιση σας, να πούμε δηλαδή πόσο σημαντική είναι η φορολόγηση για την ανάπτυξη και ότι θέλουμε να είναι αποτελεσματικό το σύστημα φορολόγησης ε, το θέματα της διαφάνειας, της ε, συνεργασίας που τίθεται, τίθεται. Όλα αυτά είναι σημαντικά και σωστά. Αλλά σε διάφορα σημεία θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αναπτυσσόμενα κράτη δεν θα προσπαθήσουν να διοχετεύσουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους και επίσης ε, στις δικές μας χώρες να προσέξουμε προκειμένου να μην, να μην δημιουργήσουμε μη ρεαλιστικά κίνητρα. Για παράδειγμα θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτές μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων τα οποία όμως δεν πρέπει να είναι αντίθετα στα ίδια συμφέροντά μας. Χαμηλή φορολόγηση, η κυκλοφορία, το round tipping που ονομάζεται στα αγγλικά, όλα αυτά που δεν αποφέρουν ουσιαστικά τίποτε στο κράτος, ε, ωφελούν μόνο τους επενδυτές και τους συνεπενδυτές από τα αναπτυσσόμενα κράτη, που τον τρόπο αυτό τελικά τα χρήματα καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αποτρέψουμε. Υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να πω ότι στο σύνολο είμαι ικανοποιημένο με τις ε, βασικές προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να είναι περίπλοκο το φορολογικό σύστημα, αλλά δεν είναι η απάντηση πάντα, δεν κρύβεται στην απλότητα. Και υποστηρίζω ασφαλώς την έκθεσή σας, Εύα. Νομίζω ότι το φορολογικό πρόβλημα αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα πολιτικής ασυνοχής. Γιατί δημιουργούμε, στο... δημιουργούμε φορολογικούς παραδείσους, οι οποίοι δεν συνάδουν με την υπόλοιπη πολιτική μας και το κράτος ε, τελικά είναι αυτό που πλήττεται. Όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα και για τη δημοκρατία, για τη δημιουργία και την οικοδόμηση ενός κοινωνικού συστήματος, το οποίο ξέρουμε ότι είναι όλο και πιο σημαντικό για την προστασία των πιο αδυνάμων. Σε περίπτωση κρίσης, επίσης, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί συνθήκες δημοκρατικού ελέγχου για να ξέρει ο κόσμος πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Νομίζω λοιπόν ότι η φορολογία περιλαμβάνει πολλά παραπάνω από τα χρήματα και κατά το παρελθόν συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στο βόρειο Εμισφαίριο ακολουθούσαμε την εξή πολιτική. Ζητούσαμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τους φορολογικούς τους συντελεστές και Νομίζω ότι αυτό πλέον πρέπει να το εγκαταλείψουμε ως σύστημα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφθοράς, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και φυσικά χρειάζονται μέτρα διαφάνειας και κατά της διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι και οι δικές μας οι εταιρείε θα περιορίζονται κατά κάποιο τρόπο να μην μπορούν να ενθαρρύνουν, να εφαρμόζουν πρακτικές διαφθοράς, γιατί αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε για να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους διαφθορά. Merci. La parole est à Madame Ο λόγος στην κυρία Γιάστραμ. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας για ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τίθεται για μένα το ερώτημα του κατά πόσο είναι σωστό να θέσουμε θέματα good governance τόσο νωρίς. Γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ενός βελτιωμένου συστήματος. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να θίξω, είναι το θέμα της άμεσης έναντι της έμεσης ε, φορολόγησης. Γιατί πολύ συχνά αναφέρεται η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιτέμενης αξίας, ο οποίος ε, θεωρώ ότι αποβαίνει βάρος των πιο φτωχών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε και το θέμα της διάστασης του φύλου, γιατί συνήθως είναι οι γυναίκες ε, αυτές που πλήττονται, οι γυναίκες οι πιο φτωχές. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν τα παιδικά ενδύματα να τα απαλλάξουμε από τη φορολογία για να υπάρχει μια ανακατανομή του πλούτου. Θα υποβληθούν και τροπολογίες. Θα καταθέσω και εγώ τροπολογίες, δεν θέλω να επισέλθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά να πω κάτι βασικό. Πρέπει να διευκρινιστούν κάποια βασικά ερωτήματα. Το θέμα των πιστών εναντί των ε, επιδοτήσεων. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα. Και τέλος να σας θέσω και μία ερώτηση. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι το θέμα της φορολογικής δήλωσης ανά χώρα. Θεωρείτε ότι πρόκειται μία προϋπόθεση εκ των ΟΚ ΑΝΕΦ. Ναι. Merci, Monsieur Goerens, vous avez la parole. Oui, euh, η έκθεσή σας είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Να υπογραμμίσω δύο ζητήματα όμως που μου φαίνονται σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικά. Κάθε χώρα χρειάζεται ένα φορολογικό σύστημα προκειμένου να χρηματοδοτεί τις δαπάνες του. Αυτό που διαπιστώνουμε στην Ευρώπη είναι ότι κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Υπάρχει μια ενδογενής ανάπτυξη που οδηγεί σε φορολογικό αβάρι που είναι διαφορετικά σε διάφορες χώρες. Πλην όμως ε, το κάθε σύστημα μπορεί να ωφελεί τους πολίτες της χώρας του. Αν όμως αντιστρέφαμε αυτά τα συστήματα, δηλαδή η Σουηδία για παράδειγμα να υιοθετούσε το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και το αντίστροφο, οι δύο χώρες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, ούτε μία ούτε η άλλη. Είναι πολύ απλό. Συνεπώς θα πρέπει να, είμαστε, να σεβόμαστε την αρχή της εταιρική σχέσης, δηλαδή ότι οι αναψώμενες χώρες θα πρέπει να ε, μπορούν να τοποθετούνται επί του, του μέλλοντός τους, να μην τους επιβάλλουμε δηλαδή τίποτα συγκεκριμένο. Η Γκάνα, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια, είχε την εξή εμπειρία. ετίθετο το, θέτημα, ε, το θέμα της ε, χορήγησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιας καινούργιας πίστοσης. Η Γκάνα ε, ήθελε ταυτόχρονα να αυξήσει τους εισαγωγικού δασμούς ε, και αυτό οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να της αρνηθεί το δάνειο. Δηλαδή της επέβαλε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη φορολογική πολιτική ε, χωρίς να προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Είναι θέμα καθαρά πολιτικό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Γκάνα απομονώθηκε και κανένα δεν την υποστήριξε. Ποιο θα μπορούσε να το κάνει μεταξύ αυτών που είναι παρόντε στην Αφρική. Η Κίνα με πουδενή. Ούτε οι ε, υπόλοιπε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει την Κάνα και εκεί μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο παράδειγμα. Ο Μπακμπό μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο που λαμβάνει η χώρα ε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας του ε, φορολογώντας ε, τις επιχείρησεις του. Στην... κανονικά αυτό θα πρέπει να γίνει με φόρους βέβαια. Okay. Αλλά στην κακτή του ελεφαντοστούν, του ελεφαντόδοντος, συμβαίνει κάτι άλλο. η κυβέρνηση δεν έχει αρκετά φορολογικά έσοδα, οπότε αυτό που κάνει είναι ε, να, τις, ε, να τους ε, ε επιβάλλει χαράτσι. όχι επειδή δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν, αλλά επειδή αυτή είναι μια πολιτική απόφαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη σχέση μας με τέτοιες χώρες. Θα πρέπει κάθε χώρα να έχει την ευθύνη των πράξεών της. Τέλος, και το αναφέρετε κι εσείς, έχουμε το εξής. Υπάρχουν άπειροι τρόποι να κοροϊδέψουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένας από αυτούς είναι να λαιλατούμε τους φυσικούς τους πόρους χωρίς να πληρώνουν δίκαιες τιμές. Ε, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ νόμιμες στη χώρα στην οποία εξάγουν το, τις πρώτες ύλες αλλά συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα στη χώρα στην οποία εξάγεται η πρώτη ύλη, παράγεται η πρώτη ύλη. και είπα και στο πλαίσιο της προηγούμενης συζήτησης πριν έρθετε, είναι, ε, είπα ότι χρειάζεται ένα ε, διαφορετικό ταβός που θα επέτρεπε να συζητήσουμε από κοινού όλα αυτά τα προβλήματα και να δούμε τι θα μπορούσε να προσφέρει ο κάθε παράγων, ο κάθε φορέας. Νομίζω ότι η ως τώρα δράση μας ε, υποσκάπτει την ανάπτυξη των ε, αξιόμενων χωρών. Χρειάζεται ένα ανταβός δύο λοιπόν, το λέω έτσι δεν έχουμε άλλο όνομα. Ε, ένα networking που θα είναι εναλλακτικό του not working, <laughs> του να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή. Χρειάζεται λοιπόν όλοι από κοινού, ε, κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρήσει, να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις. Προσπάθησα ακόμα και στην κυρία να το πω αυτό. Δεν με άκουσε βέβαια. Έχουμε δικαίωμα να μιλάμε, αλλά θα, δεν εισακόμαστε πάντοτε. Ε, αισθάνομαι λίγο αδύναμος μπροστά σε αυτή την τρομακτική πραγματικότητα. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oui, merci beaucoup, euh, Madame Jolie. Euh, cette communication a été préparée. Η ε, έκθεση, η ανακοίνωση αυτή συντάχθηκε σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα σε, ε, είχα, οι πράσινοι είχαν οργανώσει μια εκδήλωση στην οποία ε, ήταν παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ήσασταν και εσείς κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πολλά είναι τα θετικά της έκθεσης, υπάρχουν και ορισμένες αδυναμίες. Μάλλον πολλά τα θετικά τα οποία υπογραμμίζει η έκθεση και υπογραμμίζει και ορισμένε αδυναμίε τη ανακοίνωση. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα συζητήσουμε το θέμα τη ε, μείωση, για παράδειγμα, των ε, δασμολογικών εσόδων ε, εξαιτία εμπορικών συμφωνιών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όμως αυτές οι χώρες αν βασίζονται στις δασμολογικές, στα δασμολογικά τους έσοδα σημαίνει ότι δεν έχουν επαρκή φορολογική βάση. Λέτε ότι δεν κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διεύνηση αυτής της φορολογικής βάσης. Δεν το κάνουμε πράγματι γιατί προτιμούμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση για κάθε χώρα. Δηλαδή να μην πούμε χρειάζεται ε, αυτά τα μέτρα, αυτός ο φόρος για τον α ή τον β τομέα. Θέλουμε ε, προσέγγιση αναχώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές πραγματικότητες, τις εθνικές πραγματικότητες. Ορισμένες χώρες, ε, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, έχει ένα πολύ περίπλοκο φορολογικό σύστημα, αλλά υπάρχουν και χώρες που έχουν ένα πολύ αδύναμο φορολογικό σύστημα και πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να καταλήξει σε, ένα σε μια πραγματικά δίκαιη φορολογία. Η δικαιοσύνη ε, είναι ακρογωνίως λίθος αυτή μα της προσέγγιση και γι' αυτό λόγο ακολουθούμε μια προσέγγιση ανά χώρα. Μιλήσατε επίσης και για τον ΩΣΑ και για, τις, ε, ορθή, την ορθή τιμολόγηση. Γι' αυτό θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που είπατε. Ε, προκειμένου ασφαλώς να βελτιωθούμε. Ε, για το θέμα της αποτελεσματικότητας των ασιών του ΟΣΑ, για παράδειγμα, προτείνατε μια διεθνή σύμβαση για την ε, καταπολέμηση των βλαβερών φορολογικών πρακτικών. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των ουσιών του ΟΣΑ, είναι αλήθεια ότι η πρώτη φάση ήταν ο ΩΣΑ να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για τη διαφάνεια και για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων. Το δεύτερο στάδιο όμως ήταν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτών των διευθετήσεων. Δηλαδή μια διαδικασία ε, ελέγχου από ομότιμους, peer review. Η διαδικασία αυτή θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια και θα επιτρέψει να επιβεβαιωθεί πρακτικά το κατά πόσον οι αρχές διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών εφαρμόζονται στην πράξη από τα διάφορα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ. Αυτό θα επέτρεπε να εντοπιστούν οι εικονικές συμφωνίες ή συμφωνίες ευκαιρίας. Μετά, ε, μίλησατε για τη Διεθνή Σύμβαση. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας για την φορολόγηση των επιχειρήσεων που καλύπτει την καταπολέμηση των βλαβερών φορολογικών πρακτικών και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί να τον εφαρμόσουν αυτόν τον κώδικα στις τρίτες χώρες. Και αυτή η προώθηση περιλαμβάνει και ορισμένες γειτονικές χώρες της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο στόχος της ρήτρα που συστηματικά σχεδόν κατά κανόνα περιλαμβάνεται στις συμφωνίες που συνάπτουμε με τρίτες χώρες που είναι η ρήτρα της καλής ε, δημοσιονομικής διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να εξασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας, μας εγκρίνουν και εφαρμόζουν τις αρχές διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών ε, και φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα 21 διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Και νομίζουμε ότι αυτή η ρήτρα θα ικανοποιήσει τις ανησυχίες σας, θα διασκεδάσει τις ανησυχίες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, διαπιστώνω με ικανοποίηση πως υπάρχει υποστήριξη στην ιδέα αυτή στην ιδέα την οποία βρίσκεται μέσα στην έκθεση αυτή υπήρξαν προτάσεις Σνίμπερ για Στραμ ίσως να βάλουμε τα στοιχεία της καλή κυβέρνηση σαν στα συμπεράσματα αντί να πει στην αρχή, στο προήμιο να πει στα πορίσματα. Νομίζω πως τα δύο θέματα αυτά συνδέονται στενά και νομίζω πως μπορεί να πάει είτε, είτε, είτε στο ένα μέρος στο άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αφετέρου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μια απόφαση επί του θέματος αυτού δεδομένου ότι προηγουμένως παρέστην στο ΠΝΙΝΤ στο ξεκίνημα της εκθεσής όσον αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη του κνούντου ανθρώπινη ανάπτυξη. Διαπιστώνεται λοιπόν εκεί σε αυτή την έκθεση ότι υπήρξε μια ανάπτυξη συνδυασμένη μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, υγείας, εκπαίδευσης κατά 41% από το 70 μέχρι τούδε. Όταν δούμε λοιπόν την, την κατάταξη του ΚΝΟΥΤ υπάρχουν οι χώρες ερεπτυγμένες στο ΚΝΟΥΤ και όταν δούμε το 40%, 41% της ανάπτυξης αυτής που προανέφερα στα 47 έτη, θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με το ΑΕΠ, στο ΑΕΠ των τελευταίων αυτών 40 ετών και το οποίο είναι της τάξης του 50%. Αυτός είναι ένας λόγος επιπλέον για ε, του δείγματος ότι δεν υπάρχουν έσοδα φορολογικά των αναπτυσσομένων χωρών για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιες εκείνες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην οικονομική και εκπαιδευτική λοιπά αναπτύξεις. Για πολύ χρονικό διάστημα εγκαταλείψαμε ε, να εγκαταλείψουμε το σύστημα και υπάρχει ένα δημοσιονομικό σύστημα το οποίο, σύστημα το οποίο είναι βλαβερό και το οποίο οι συμβάσει του ΟΣΑ είναι μη αποτελεσματικέ. Γιατί, διότι θα πρέπει να δημιουργούν, να, δει, συγγνώμη, να ζητηθούν οι πληροφορίε εκείνε, αλλά, αλλά δεν γνωρίζουν πραγματικότητα τα χρήματα αυτά βρίσκονται σε, σε δημοσιονομικούς παραδείσους και άρα η πληροφορία δεν έρχεται. Επίδειξη αυτού του λεχθέντος είναι η συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και των χρόνων αυτών και υπάρχει και το μοντέλο του ΟΣΑ αυτό χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από 10 φορές. Είναι μια τεράστια εργασία, εργασία η οποία πρέπει να γίνει για διμερές συμβάσεις, για διμερείς συμβάσεις συγγνώμη, πρέπει να γίνουν. Είναι λοιπόν σημαντικό όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλάβει τις ευθύνες υπό την σκοπιά της ανάπτυξης διότι υπάρχει τεράστια υποκρισία και ακόμη οι δυνατότητες να μην πληρώνονται φόροι σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, νομίζω πως με ευχαρίστηθη η θεάθη εκ μέρους των επιχειρήσεων που εργάζονταν εκεί και αυτό δημιούργησε περαιτέρω δυσκολίες μεταξύ του. Ευχαριστώ λοιπόν που, ε, που καταθέσατε τις τροπολογίες σας. Πριν από τις 16 Νοεμβρίου, τόσο και θα γίνει στις 18 Γενάρη του 2011 η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. θα τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ είμαι η συγγήτρια, διότι ούτε ήθελε να το αναλάβει, το ανέλαβα εγώ, σαν πρόεδρος. Μου δίδω το λόγο και μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρίς κείμενο, επαναλαμβάνω, η επόμενη έκθεση μου θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου και η προθεσμία θα είναι μέχρι και πρωί μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια τεχνική προσαρμογή που γίνεται σε θέματα συνεργασίας και το οποίο προβλέπεται από τη συνθήκη της από την εισαγωγή ενισχύει της ε, συνθήκης της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πρέπει να άπτεται αυτού του θέματος και ε, θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο στο όνομα της ΕΕ αλλά επίσημα θα πρέπει να κοινοποιείται επισήμω στη Νότια Αφρική και από το Γενάριο του 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποκαθιστά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα επισήμως και ό,τι προκύπτουν από τη συμφωνία αυτή και ιδιαίτερα το άρθρο 217 όσον αφορά την λειτουργία 17 ε, και σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 βλέπετε, προβλέπετε ότι όλα αυτά μπορούν να τεθούν λειτουργία μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση που λοιπόν θα εξεταξεί στις 9 Δεκεμβρίου συστήνει εξ ονόμου της Επιτροπής μας το Κοινοβούλιο να δεχθεί ο σώμα πλέον την πρόταση την οποία έχουμε αναχείρας. Όπως βλέπετε αυτό προκύπτει από το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας και ιδιαίτερα από το 218 και ότι σύμφωνα με αυτό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να εισαχθούν τροπολογίες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συστήσουμε προς την Ολομέλεια την αποδοχή ή την απόρριψη, τίποτα άλλο. Συνεπώς, όσον αφορά τη διαδικασία λοιπόν, καθώς επίσης και την διαβούλευση με άλλες επιτροπή, η ίντα είναι αυτή η οποία θα δώσει τη γνώμη της, ενώ επί της ουσίας είμαστε αρμόδια εμείς η Επιτροπή που θα πρέπει. Θα πρέπει οπωσδήποτε βεβαίω να περάσει αυτό από το σώμα στην ολομέλειά του για να μπορέσει να εισαχθεί αυτή η αναθεωρημένη συμφωνία. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 26 Γενάρη του 2011 και οι τροπολογίες που θα τεθούν είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου παραλαμβάνω. Εδώ τι είχα να πω. Αυτά. Έχετε το λόγο εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια κλπ. Λαμπρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Πέρα στη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί στις 10 και οι θα συνέλθουν στι 9 και 30 παρακαλώ σημειώσατε 9 και 30 στην ίδια αίθουσα. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα σας.